Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place puisque... Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, διότι μόλις κατέφτασαν οι ομιλητές μας για το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Σα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή μας συνεδρίαση στο σημείο 14. Περνάμε λοιπόν θα γίνει ένας απολογισμός των συμφωνιών που συνήφθησαν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και ο κύριος Αρμίντα Ντασίλβα, διευθυντής αμπεαρμόδιος για την απασχόληση ε, και τον κοινωνικό διάλογο στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ απασχόληση είναι μαζί μας σήμερα. Νομίζω ότι έχετε λάβει ένα θετικό φάκελο. Το βασικό διακύβημα για την ανταλλαγή απόψε είναι η παρακολούθηση της συνέχειας που εδόθη στη συμφωνία που συνυπέγραψαν οι κοινωνικοί εταίροι. Ε, κύριε Γενική Διευθυντά, θα σας δώσω το λόγο για μια παρέμβαση δεκάλεπτη ε, κατά προτίμηση. Σας ακούμε. Καλημέρα. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω που προσκαλέσατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ως προς με τους κοινωνικούς εταίρους. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να προάγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον κοινωνικό διάλογο και βάσει του άρθρου 155 της συνθήκης Βλέπουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι έχουν επίσης την αρμοδιότητα να διαπραγματευτούν ε, συμφωνίες για την κοινωνική πολιτική και να ζητήσουν ε, την εφαρμογή τους μέσω οδηγιών του Συμβουλίου. Η διαδικασία αυτή δεν έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολλές φορές μέχρι στιγμή, αλλά ε, και σε κλαδικό επίπεδο και σε επίπεδο βιομηχανίας υπάρχει προηγούμενο. Έχουμε οδηγίες στο κοινωνικό πεδίο Παραδείγματο χάρη οδηγία για τη γονική άδεια, ε, για την εργασία μερικού χρόνου, για τις ε, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την ε, υγεία και την ασφάλεια στη χώρο εργασίας και τα ωράρια εργασίας. Το 2012 ο κλαδικός κοινωνικός διάλογος οδήγησε και στην υπογραφή δύο συμφωνιών και εφαρμογή τους μέσω της, κοινωνικής, της ενωσιακής νομοθεσίας ζητήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε παραδείγματος χάρη για τις εσωτερικές Πλωτού πλωτούς οδούς και για την ε, υγεία και την ασφάλεια στον τομέα των κομμωτηρίων ε, ε, διέπονται από δύο οδηγίες που προκύπτουν από τις συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους. Κλαδική συμφωνία επίσης για τι εργασιακέ συνθήκες στην αλληλεία, στη θάλασσα. Και ο στόχο είναι πάλι να χρησιμοποιήσουμε την οδό τη οδηγία του Συμβουλίου για την εφαρμογή. Αναμένεται επίσης για το χώρο εργασίας, για την αναθεώρηση οδηγίας για το χρόνο εργασίας, αναμένεται λοιπόν η περάτωση των διαπραγματεύσεων στο τέλος του 2012 και αναμένεται να ζητήσουν εφαρμογή μέσω της ε, οδηγίας. Ε, οι διαπραγματεύσεις ε, άρχισαν μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι όροι εφαρμογής αυτών των διατάξεων της συνθήκης διευκρινίστηκαν σε διαδοχικές ανακοινώσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής η τελευταία χρονολογία το 2012. Ε, δύο. Ε, η, το Συμβούλιο δεν δύναται να ε, τροποποιήσει αυτές τις συμφωνίες. Μπορεί να δεχτεί ή όχι να καταστήσει δεσμευτικές ε, τις διατάξεις της συμφωνίας επί τη βάση μιας πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενημερώνεται το Κοινοβούλιο για τη διαδικασία, δεν έχει όμως ε, κανένα άμεσο ρόλο. Η διαδικασία κατοχυρώνει πλήρω το δικαίωμα πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν υποχρεούται να καταθέσει πρόταση νομοθετικού περιεχομένου στο Συμβούλιο. Όμω, όπω προβλέπεται ρητά μέσα στι ε, διαδοχικέ ανακοινώσει που προανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τη δέσμευση να αποτιμήσει το περιεχόμενο τη συμφωνία και αν δεν ε, προτείνει την εφαρμογή της μέσω και νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμή, οφείλει να ενημερώσει τους κοινωνικούς εταίρους ε, για την αιτιολόγηση τη απόφαση τη, Η αποτίμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επικεντρώνεται στην νομιμότητα τη συμφωνία ε, του τέστην ε, αν συμμορφώνεται με, το, με την κείμενη νομοθεσία, τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων μερών και τι επιπτώσει επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε περίπτωση συμφωνιών ε, που δεν προέρχονται από αυτή τη διαδικασία διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για τα κομμωτήρια και την εσωτερική ναυσιπλοεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να εκτιμήσει την ε, δυνατότητα του ενδεχόμενου ανάληψης σε δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τώρα από αυτές τις οδηγίες για την υγεία, η οδηγία για την ε, υγεία και την ασφάλεια στα κομμωτήρια δέχθηκε επικρίσει, ε, κυρίως από πλευράς κάποιων κρατών μελών. Αυτή η συμφωνία βασίζεται ε, σε μακρά εργασία των ε, κοινωνικών εταίρων που συνέλεξαν επιστημονικά στοιχεία σε σχέση με τους ειδικού κινδύνους ε, σε αυτόν τον τομέα. Παραδείγματο χάρη αλλεργίες στο αναπνευστικό σύστημα ή χαμηλή ηλικία συνταξιοδότηση που απαιτείται σε αυτόν τον τομέα, καθώς και βέλτιστες προακτικές από την εφαρμογή της νομοθεσίας σε κάποια κράτη-μέλη. Ποιες είναι οι επικρίσεις που λάβαμε. Δεν αμφισβήτη η οι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία σε αυτόν τον κλάδο, όμω, η προσέγγιση της κλαδική προσέγγιση στην νομοθεσία ε, για, στον τομέα τη υγεία και τη ασφάλεια στον χώρο εργασία τίθεται να αμφιβόλο. Ζητήθηκε μερική αναθεώρηση τη οδηγία, διότι θεωρείται ορισμένε φορέ υπερβολικά διεξοδική και ότι δεν συνάδει με τι αρχέ επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Μάλιστα. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίω από τη ΓΔ Απασχόληση, ανέλαβαν τη δέσμευση να εξετάσουν τι σε ήδη κατατεθεί σε συμφωνίες καθώς οι εκείνες που αναμένονται επί τη βάση των κοινών κανόνων. Αυτό τι σημαίνει ανάλυση της εκπροσωπευτικότητας, ε, νομική συμμόρφωση, επιπτώσεις επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς ε, και ε, ανάλυση της, των νέων ευκαιριών. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε του κανόνες ενώ διαρκεί το παιχνίδι ως προς την αξιολόγηση των επιπτώσεων των συμπεφωνημένων λύσεων θα βασιστούμε σε μελέτες κόστους γνωστούς σε τώρα ε, ξεκινούμε. Οι μελέτες αντικτύπου θα ε, δημοσιευθούν. Η απόφαση του αν θα κατατεθούν ή όχι προς έγκριση στο Συμβούλιο αυτές οι συμφωνίες ε, θα βασιστεί επί αυτών των αξιολογήσεων που αναμένουμε να ολοκληρωθούν μέχρι το πρώτο ήμιση του 2013. Αυτή είναι η άμεση δράση που ε, θα να αναλάβουμε για να αντεπεξέλθουμε στην κατάσταση. Τώρα, πιο μακροπρόθεσμα και για το μέλλον, να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μία ανάγκη να αναλύσουμε διεξοδικά τις πρακτικές εφαρμογής του Άρθρου 115 τη της συνθήκης ε, ε, υπό το φως των αρχών και των πρακτικών ε, του θεματολογίου της ευφιέστερης νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. Επ' αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όμως διατηρεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της και πρέπει να μεριμνά ούτως ώστε όλες τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου να συνάδουν με τις αρχές της ευφιούς νομοθεσίας, δηλαδή αναλογικές, εναργώς διατυπωμένες και στόχευμένες Επίση Επίσης πρέπει να αντιλήσουμε διδάγματα από την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από τα προηγούμενα έτη με την εφαρμογή ε, ενός αριθμού ε, συμφωνιών ε, με τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα εξετάζουμε το ενδεχόμενο επικαιροποίηση και διευκρίνηση των όρων εφαρμογής των συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους. Η τελευταία ανακοίνωση που είχαμε σχετικά είναι από το 2002, όπως σας είπα, πριν προδεκαετίας. Άρα Εξού μάλλον και ανάγκη επικαιροποίηση ε, υποδοφός το της ε, εμπειρίας που έχουμε πλέον και να διευκρινίσουμε στου κοινωνικούς εταίρους ότι όπως και στην περίπτωση άλλων νομοθετημάτων θα πρέπει να καταδεικνύεται ε, σαφέστατα η, σαφέστατα οι θετικέ επιπτώσεις αυτών των συμφωνιών. σε ευχαριστούμε. Η η ε, Κοινωνική Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας ε, υπέδειξαν ότι υπάρχουν ατέλειες και λήψεις ως προς το σεβασμό των αρχών του κοινωνικού διαλόγου, ως προς τις ε, συλλογικές διαπραγματεύσεις και το ρόλο αυτών των κοινωνικών ετών, οπότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει ένας απολογισμός. Έχω διάφορες ερωτήσεις, θα αφήσω όμως πρώτα τους συναδέλφους μου να παρέμβουν και Ρωτώ ποιο θα ήθελε το λόγο παρακαλώ για αυτό το θέμα. Σέρκας. Φάρμπρ, θέλετε το λόγο. Όχι. Σέρκας, παρακαλώ. Sí, señora presidenta. Este es Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα, κύριε Πρόεδρε, που όπου δεν θα καταλήξουμε σε κάτι σήμερα διότι υπάρχει μια διένεξη σημαντική εδώ. Έχουν, δεν έχουμε συμφωνίες συγκεκριμένες. Υπάρχουν πολλοί δομείς. Εδώ μιλάμε για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε διάλογο και εδώ έχουμε ένα άρθρο που αναφέρεται σε αυτό ότι πρέπει να συνεχιστεί αν υπάρχει επιθυμία αλλά θα πρέπει να καταλήξουμε στις συμβάσεις συλλογική. Ό,τι γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να γίνει, είναι συμβατό με τις χώρες μέλη. Θα περάσουμε σε μια απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, του, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συγγνώμη. Εδώ είναι πολύ σαφές ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει ότι αυτό επιθυμεί πέρα από κάθε λογική με βάση το κοινωνικό διάλογο. Η Επιτροπή αυτό που είναι εξαφέσαν είναι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τη συνθήκη. Τι είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εγγυητής της σύμβασης. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα όπως και στο παρελθόν. θα πρέπει να ισχύουν, να περάσουν σε ισχύ οι όποιες συμφωνίες έχουν συναυθεί. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι καταργηθεί η δυνατότητα για τους κοινωνικούς να ε, καθορίσουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο δουλεύουν. Θα πρέπει να το δούμε αυτό αυτό που βλέπουμε στη διουσία, αυτό που γίνεται τώρα. Είναι μια επίθεση στο, ε, θα λέγαμε, συνταγματικό βάθρο της Ευρώπης. Έχουμε αυξηθεί, περάσαμε από το 8, 10 και 15 τώρα μέλη. Και αυτό που γίνεται, τι γίνεται. Γίνονται διάφορες δραστηριότητες λόμπι που επηρεάζουν τις διαδικασίες. Θα πρέπει να αναγνωριστεί η ε, η χάρτα που ισχύει για τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν πρέπει να καταστρατηγηθεί κάτι τέτοιο. Και θα πρέπει φυσικά εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να εφαρμόσει τις αρμοδιότητές της. Σίγουρα η Επιτροπή θα έχει την υποστήριξη όλης της ομάδας μας για να ολοκληρώσει το καθήκον της. Να μην τρομάξει, να μην υποχωρήσει. Είναι ένα επικίνδυνο ε, σημείο τώρα. Ηνωμένο, Βασίλειο. Πάντοτε πρώτο. Μετά έχουμε Πολωνία, Στονία, οι κάτω χώρες, Σουηδία, Σλοβανία και, η Σλοβενία και η Κροατία. Τι ακριβώ γίνεται. Δεν αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι χώρες. Είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν υπάρξουν κάποιοι άλλοι. Παρακαλώ. Ο κύριος Φάμπρα. Mám stejný názor a na přítomného zástupce mám dotaz. Mluvil o tom, že... Ναι, συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν μόλις και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι την Επιτροπή. Μίλησε η Κομισιόν για μια νέα οδηγία για την εργασία Ξέρουμε τι έχει συμβεί. Θα ήθελα να μου πείτε τι θέλετε να συμπεριλάβετε σε αυτή την οδηγία. Υπάρχουν. Άλλοι που ζητούν το λόγο. Ε, ε, ο κύριος Ντασίλβα, ε, ε, λοιπόν, δεν έχω μπροστά μου την ημερομηνία αυτής της πλέον γνωστής επιστολής, της διαβόητης επιστολής των εκείνων που απορρίπτουν τον, τον αντιστασιακό προς τον κοινωνικό διάλογο. Αυτή η επιστολή εστάλει, όπως γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρω σε ποια ημερομηνία. Ε, θα ήθελα να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία με τη συμφωνία για την εσωτερική ναυσιπλοεία όπως και για τους κομμωτές διότι για την εσωτερική ναυσιπλοεία Έχω την εντύπωση ότι δεν σας εμπόδισε αυτό να προχωρήσετε. Η συμφωνία έγινε 15 Φεβρουαρίου. Ε, τι, Φεβρουαρίου, τι προβλέπετε λοιπόν Τώρα όσον αφορά την συμφωνία για τους κομμότες της 26 Απριλίου μας είπατε ότι ξεκινήσατε μια μελέτη επιπτώσεων. Πότε το αποφασίσατε αυτό, ποιος θα την πραγματοποιήσει αυτή τη μελέτη έτσι, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθούνται πάντα. Είπατε ότι όσον αφορά τις συμφωνίες θα πρέπει να μελετήσετε μια σειρά κριτηρίων ώστε να επαληθεύσετε κατά πόσο μπορούν να ε, καταλήξουν νομοθεσίε. Τώρα στο θέμα της συμφωνίας για τον τομέα της κομματικής ε, πώς ε, καλύπτονται τα κριτήρια που πρέπει να μελετήσετε. Αναφέρατε για παράδειγμα την αντιπροσωπευτικότητα. Μπορείτε να τσεκάρετε δηλαδή το σύνολο των κριτηρίων, το σύνολο των συνθήκων που μπορείτε να μετατρέψετε σε συμφωνία. Που μπορείτε να μετατρέψετε από συμφωνία σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση για την οποία θα επιθυμούσα να μου δώσετε μια απάντηση. Euh, ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας ξεκινώντας από την ημερομηνία της επιστολής που λάβαμε από τον ε, ε, Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων της Ολλανδίας και από εκπρόσωπο ε, αντιπροσώπειες 9 κρατών μελών και από την Κροατία 25 Οκτωβρίου του 2012. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή προχωράμε ε, για τη συμφωνία για την εσωτερική ναυσιπλοεία και για τους κομμωτές με τον ίδιο τρόπο. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτές τις μελέτες αρχές Σεπτεμβρίου Όταν ε, κατέστη, προφανές ότι δεν μπορούσαμε ε, επειδή χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία πληροφοριών ανάλυσης από τους κοινωνικούς εταίρους ε, που θα μας επέτρεπαν να αξιολογήσουμε τη διαφορά μεταξύ των κανόνων που ήδη έχουν εγκριθεί και των κανόνων που ουσιαστικά εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη-μέλη καθώς και στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε τις οικονομικές κοινωνικές επιπτώσεις για τις συνθήκες εργασίας από τις νέες διατάξεις σε σχέση με αυτό που υπάρχει ήδη. Εμείς ε, ζητήσαμε αυτά τα στοιχεία από τους κοινωνικούς εταίρους, κυρίως στην ιστορική πλοία και δεν καταφέραμε να λάβουμε καμία πληροφορία από αυτές που χρειαζόμαστε και εκεί αποφασίσαμε να ε, πραγματοποιήσουμε μελέτες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να καταλάβουμε καλύτερα το αντίκτυπο των νέων διατάξεων στις συνθήκες εργασίας του τομέα. Δύο μελέτες λοιπόν, οι οποίες θα διεξαχθούν από εξωτερικούς αναδόχους, έχουν ήδη ξεκινήσει. Μία μελέτη για την εσωτερική ναυσιπλοεία, μία άλλη για τους κομμωτές. Μελέτες που κυρίως αναμένουμε να μας δώσουν απαντήσεις εν τέλει σε σχέση με τη διαφορά κόστους και ωφελών από οικονομική και κοινωνική άποψη. Το θέμα της αντιπροσωπευτικότητας αναλύεται σε μελέτες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας ε, στο Δουβλίνο, την Eurofound, είναι διαθέσιμες αυτές οι μελέτες και μας επιτρέπουν να συμμετήσουμε μια εικόνα του βαθμού αντιπροσώπευσης ε, των ε, υπογραφών των δύο συμφωνιών. Τώρα, όσον αφορά τα κριτήρια συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αυτή είναι μια εργασία που γίνεται με δική μα μέρημνα. Εξάλλου, έχουμε ήδη ξεκινήσει αυτή την εργασία εδώ και αρκετό καιρό. Έχουμε προχωρήσει δηλαδή αρκετά αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να εκτιμήσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις και για αυτό πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ των πραγμάτων που υπάρχουν σε διάφορα κρατή-μέλη και των πραγμάτων που προτείνονται. Προφανώς, όπως και για την αξιολόγηση αντικτύπου, όπως και για την έξυπνη νομοθεσία, αυτές είναι διαδικασίες που βελτιώνονται. Σήμερα πιστεύω οι δικές μας νομοθετικές προτάσεις βασίζονται καλύτερα σε πραγματικά γεγονότα από ό,τι συνέβαινε πριν από 10 χρόνια. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τις ίδιες αρχές και στις συμφωνίες που λαμβάνουμε από τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να τηρεί τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου. Αλλά αυτή τη στιγμή οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν από την Κομισιόν να παρουσιάσει μια νομοθετική πρόταση στο Συμβούλιο η Κομισιόν πρέπει να αξιολογήσει επίσης και την ποιότητα αυτής της πρότασης. Η Κομισιόν λοιπόν δεν είναι ένα ε, ε, κουτί αλληλογραφίας ε, διατηρεί ένα δικαίωμα πρωτοβουλία το οποίο ασκεί σε αυτή την περίπτωση όπως θα κάνει και για οποιοδήποτε άλλη πρόταση νομοθετήματος. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν από την Κομισιόν στοιχεία, πληροφορίες που θα τους επιτρέπει που να γνωρίζουν ποιε θα είναι οι επιπτώσει τη νομοθεσία που θα κληθούν να εφαρμόσουν. Έλαβε λοιπόν αυτή την επιστολή η Κομισιόν. Πρόκειται για μια τοποθέτηση ορισμένων κρατών μελών. Αυτό δεν μετακινεί την Κομισιόν από τη θέση τη. Είχε αποφασίσει να ξεκινήσει αυτέ τι μελέτε πριν λάβει την επιστολή από τα κράτη-μέλη. Ε, τέθη επίση το ερώτημα τη αναθεώρηση τη οδηγία τις οδηγίες ε, περί χρόνου εργασίας. Αναμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όχι και μέσα στις επόμενες μέρες, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, των κοινωνικών εταίρων, σε διεπαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή το Business Europe, ε, CP, WATME και, σε, και ΕΟΚΕ έχουν ξεκινήσει αυτές τις διαπραγματεύσεις στα τέλη του 2011 και έχουν δεσμευτεί να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών μέσα στις επόμενες εβδομάδες ή μάλιστα και ημέρες. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα, συνεπώς δεν μας είναι δυνατό αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε αυτά τα αποτελέσματα, η Κομισιόν θα αναλύσει. Λοιπόν και τα αποτελέσματα αυτών των διαπραγματεύσεων και έχει την πρόθεση επίσης ε, να παρουσιάσει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με κάποια σχετική ανάλυση και αξιολόγηση στο Συμβούλιο, ε, συγγνώμη, στους ε, επιτρόπους, ώστε ε, το κολέγιο των επιτρόπων να μπορέσει να προχωρήσει, να λάβει τις αποφάσεις που θέλει. Αλεξάνδρο, η απάντηση του κυρίου Σίλβα θέτει νέα ερωτήματα όσον αφορά εμένα, διότι προφανώς η Κομισιόν δεν είναι απλά ένα ταχυδρομικό κουτί. Κανείς ε, δεν θέλει να αφαιρέσει την ικανότητα ανάλυσης από την Κομισιόν, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ανάλυση της ποιότητας, αλλά και ανάλυση των αρχών που υπάρχουν στην επιστολή και στις συνθήκες και του ρόλου που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω εγώ είναι κατά πόσο η διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτές τις δύο περιπτώσεις είναι ίδια με εκείνη που ακολουθούμε ε, παραδοσιακά. Δεν είναι να αναφερόμαστε σε μια επιστολή από τα κράτη-μέλη, διότι πριν από την επιστολή, πριν σταλεί αυτή η επιστολή, είχε τοποθετηθεί η Ομοσπονδία Κόμματων του Ηνωμένου Βασιλείου με μια σειρά δηλώσεων και λόμπινγκ και δραστηριότητε εξάσκηση πίεση κατά δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά των κοινωνικών εταίρων. Αλλά υπάρχει ακόμη και αυτό που συμβαίνει στι κατοχώρε. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε ενώπιον συντονισμένης πίεσης από ορισμένου εργοδότες βλέπουμε να ασκείται τεράστια πίεση ώστε να υπονομεύσει αυτό που έχει επιτύχει η συνθήκη ελεύθερα μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές οι αρχές λοιπόν που αναφέρονται στην επιστολή, την οποία μας αναφέρει ο κ. Σίλβα, οδήγησε σε μια ανάλυση, σε μια αξιολόγηση που διεξάγεται διαφορετικά σε σχέση με το τι γίνεται στο παρελθόν. Ακολουθώντας τη... Ακολουθούμε τις ίδιες διαδικασίες ή και η Κομισιόν ε, υπόκειται σε αυτή την πίεση αυτών των οργανισμών που την αναγκάζουν να αλλάξει τις διαδικασίες της. Σας ευχαριστώ. Γιατί το Ίδρυμα που έχει εξετάσει το θέμα. Έχουμε πάρει αποτελέσματα για αυτή την αξιολόγηση. Μήπως θα μπορούσατε να μας τα ανακοινώσετε για τη συμβατότητα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, νομίζω ότι έχει γίνει κάτι και σε αυτό. Θα μπορούσατε και γι' αυτό να μας ενημερώσετε. Τη στιγμή που έχουμε και μια συμφωνία η οποία έχει επιτευχθεί από το Φλεβάρι Επιτρέψτε μου επιπλέον μια γενική παρατήρηση. Δεν έχει να κάνει με τις ικανότητές σας να απαντήσετε, αλλά για το διάλογο, το δημόσιο που έχουμε. Υπάρχει στην Επιτροπή, υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο να γίνεται στην πρακτική της όταν είχαμε το θέμα της εφαρμογής του six-pack. Απ' τη μια θα μου πείτε φυσικά αυτό ήταν για να σωθεί το ευρώ. Τώρα έχουμε τον διάλογο τον κοινωνικό. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα ίσως. Η τελευταία ερώτηση. Λέτε ότι δεν είναι ένα γραμματοκιβώτιο η Επιτροπή. Προσπαθεί να κάνει το έργο της. Θα ήθελα να πω στο κοινωνικό τώρα αυτό θέμα που συζητάμε, τα κοινωνικά μάλλον θέματα, δημιουργούν το ερώτημα αν μια τέτοια πρωτοβουλία και αν εσείς δεν είσαστε ένα γραμματοκιβώτιο σε σχέση με τους κοινωνικούς εταίρες τι θα κάνετε με αυτό το γράμμα τέλος πάντων διότι με αυτό καταστρατηγείται το δικό σας μονοπόλιο της ε, πρωτοβουλία. Θέλετε να διατηρήσετε το πεδίο ε, κινήσεώς σας. Ε, αλλά ποια είναι η βασική πρόθεσή σας, περιμένοντας φυσικά και τα αποτελέσματα για όλες τις μελέτες που έχετε ξεκινήσει. Υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα με τις χώρες μέλη που καταστρατηγεί το δικό σας μονοπόλιο όσον αφορά την πρωτοβουλία. Και άλλο ερώτημα θα είχα, αλλά δεν θέλω να σας ε, ε, κουράσω με αυτά, να μην παρατείνω πολύ το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης. Σας ευχαριστώ και θα θέλω να απαντήσετε σε αυτές, ε, εκ νέου σε αυτές τις ερωτήσεις. Κι άλλη μια, κι άλλη μια. Για το χρόνο εργασίας, στην οδηγία που αναφέρατε βλέπουμε δεν, είναι η ίδια, δεν εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία, αλλά από την αρχή αυτής της ε, κοινοβουλευτικής διαδικασίας, θα ήθελα να πω, είδαμε ότι είναι οι κοινωνικοί εταίροι αυτοί που θα πρέπει να βρουν μια συμφωνία, να πετύχουν μια συμφωνία. Και εμεί είπαμε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, αν υπάρχει, φυσικά θα το υποστηρίξει η Επιτροπή, αλλά αν δεν υπετυχθεί κάτι τέτοιο, θα, θα ξεκινήσει μια. θα ασκήσει το δικαίωμά τη για την πρωτοβουλία η Επιτροπή. Τώρα, αν υπάρχει μια συμφωνία ε, ή δεν υπάρχει τέλο πάντων μια συμφωνία ανάμεσα στου κοινωνικού εταίρου, οι χώρε μέλη μπορούν να σα στείλουν πάλι μια επιστολή. Θα βρεθούμε σε ένα διέξοδο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και εδώ έχουμε να κάνουμε το θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το θέμα της ανταγωνιστικότητας, Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω επεξηγώντα ένα σημείο. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς για να αξιολογήσουμε τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων είναι τα ίδια σήμερα όπω ήταν ανέκαθεν. όπω είπε ο κύριο Σέρκα, δηλαδή αναλύουμε την εκπροσώπηση τη συμμόρφωση με το κοινοτικό κεκτημένο ανάλυση επιπτώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο πλαίσιο, στην περίπτωση μάλλον συμφωνιών που έχουν συναυθεί με πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων χωρίς διαβούλευση με την Επιτροπή ε, με ανάλυση της σκοπιμότητας ε, και του ωφέλους της συμφωνίας. Ε, Αναφέρθηκα σε εκείνη την ανακοίνωση το, σε δεκαετίες του 1990 και του 2002. Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Ε, εκεί που έχουμε γίνει πιο απαιτητικοί είναι ουσιαστικά η ποσοτική βάση βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία της αναλυσής μας. Ιστορικά παρατηρούμε ότι έχουν εξελιχθεί οι προτάσεις της Κομισιόν σήμερα. Οποιαδήποτε πρόταση της Κομισιόν συνοδεύεται με μια εκτίμηση αντικτύπου βάσει ποσοτικών κριτηρίων. Υπάρχει μια ιστορική εξέλιξη και θέλουμε εμείς να εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές ώστε να θεμελιώνουμε καλύτερα τις αναλύσεις μας βάσει στα ίδια κριτήρια όπως χρησιμοποιούνται στο παρελθόν. Αυτό δεν αλλάζει. Όπως είπα, το επαναλαμβάνω, η, η απόφαση του να βασιζόμαστε σε στοιχεία πιο ρεαλιστικά τα οποία μας παρέχουν οι κοινωνικοί εταίροι είναι μια απόφαση που λάβαμε πριν την επιστολή των κρατών ε, των κοινωνικών εταίρων. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η Κομισιόν λαμβάνει επιστολές από τους κοινωνικούς εταίρους ή από τα κράτη-μέλη είτε από διάφορα κινήματα οργανισμούς, ενώσεις ε, διάφορες ε, γνωρίζοντα ότι ετοιμάζει μια νομοθετική πρωτοβουλία η Κομισιόν και έτσι ασκούν πίεση όπως είπατε στην Κομισιόν για να κάνει το ένα ή το άλλο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτή η επιστολή φυσικά χρειάζεται να απαντηθεί αλλά ε, αυτή η επιστολή δεν πρόκειται να επηρεάσει την εφαρμογή των κριτηρίων από την Κομισιόν Θα στείλουμε λοιπόν απάντηση στην επιστολή αυτή, αλλά δεν είναι παρά μία επιστολή μεταξύ άλλων που απευθύνουν διάφοροι στην Κομισιόν ε, για να κατευθύνουν την Κομισιόν προς να κατεύθυνση ή άλλη. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για το χρόνο εργασία και τι σχετικέ διαπραγματεύσει, εκεί θα εφαρμόσουμε τα ίδια κριτήρια. Είναι ε, προφανέ. Δεν υπάρχει λόγο να μην τα εφαρμόσουμε. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διεξάγονται, τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιοποιηθούν ταυτόχρονα. Δηλαδή η ανάλυση εκπροσώπησης δεν θα δημοσιοποιηθεί πριν την ανάλυση κόστος όλα θα δημοσιοποιηθούν ταυτόχρονα. Πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας όσον αφορά την εκπροσώπηση μας κάνουν να πιστεύουμε ότι πληρούνται τα κριτήρια και στις δύο περιπτώσεις προς το παρόν. Δηλαδή και στην περίπτωση των κομματών και στην περίπτωση της εσωτερικής ναυσιπλοείας. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών ε, θα λάβει χώρο, χώρα μαζί με την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης. Ναι, ευχαριστώ. Εν συντομία, κυρία Πρόεδρε θεωρώ υποχρέωσή μου να πω στον κύριο Σίλβα ότι ε, στη, η δική μου ομάδα δεν θα ακολουθήσει αυτή την οδό. Δηλαδή η υποβάθμιση της αξίας ε, της επιστολής ε, αυτών των κρατών μελών σαν να είναι μια οποιαδήποτε επιστολή που λαμβάνει από την κοινωνία των πολιτών. Εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη μιλούν στο Συμβούλιο και θα πρέπει να μιλήσουν αφού έχουν στα χέρια τους την πρόταση της Επιτροπής. Αλλά δεν θα πρέπει να προσπαθούν να επηρεάζουν ή να απέχουν από το να επηρεάζουν την Κομισιόν από, την ελεύθερη, από τον ελεύθερο ορισμό των κριτηρίων. Δεν είναι λοιπόν ανώδυνο το ζήτημα αυτό. Είναι σημαντικό ως προς το περιεχόμενο και μου φαίνεται περίεργο που η Κομισιόν ε, δεν είναι θεματοφύλακα των συνθηκών και ενώπιον του Συμβουλίου ε, Πρόεδρος. Ε, αυτό. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο στη συζήτηση με τον κύριο Σίλβε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να συμμετάσχετε στη σημερινή μας συζήτηση. και κάποια μέλη της Επιτροπής ή εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων ε, θα μπορούσαν να αντλήσουν τα δικά τους διδάγματα από αυτή την ανταλλαγή απόψε. Ολοκληρώνεται έτσι αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και πάμε πίσω στο χρόνο με την ε, χρονομηχανή και επιστρέφουμε στο σημείο που έπρεπε να είχαμε εξετάσει κανονικά εχθές, ε, δηλαδή το σημείο 11. Ένα λεπτάκι να δω πώς το λένε στα γαλλικά προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση που συνέταξε η Νάντια Χίρς Ε, προς κατάθεση στην Επιτροπή ε, Προσωπικών Ελευθεριών ε, και ο Γιάνν Άλμπρεχτ από τους Πράσινους είναι ο σκιώδης εισηγητής από την καθήλυνα αρμόδια Επίτροπη. Παρακαλώ κυρία Χίρης, σας ακούμε για την παρουσίαση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος για την προστασία των δεδομένων και σαν Επιτροπή για την Απασχόληση έχουμε τη δυνατότητα να, δώσουμε, να κάνουμε την ομοδότησή μας. Θα προσπαθήσουμε κατά με να επικεντρωθούμε στο άρθρο 82. Υπάρχει πολλή συζήτηση και για άλλες, και άλλα άρθρα, κυρίως στην ΛΙΜΠΕ. Για το άρθρο λοιπόν που ανέφερα το 82 εδώ είναι το βάρος μας. Είχαμε συνάντηση με σκιώδη CT να δούμε τη μέθοδο που θα ακολουθήσουμε και συμφωνήσαμε γενικές γραμμές να δώσουμε έμφαση στο άρθρο 82 που θα μας δώσει τη δυνατότητα να ακουστεί η φωνή μας. Η συζήτηση θα συνεχιστεί στα πλαίσια της Επιτροπής. Μέχρι στιγμής το άρθρο 82 που έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια της απασχόλησης των εργαζομένων. Ήταν ένα στοιχειώδης ε, κανονισμός και είχε προβλεφθεί να γίνουν κάποιες συλλογματικές ρυθμίσεις. Στις διάφορες χώρες μέλη έχουμε διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά την προστασία δεδομένων των εργαζομένων και καταρχήν σε πρώτη φάση είχαμε να κάνουμε την αλλαγή της διατύπωσης. Άλλες χώρες που έχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας να το διατηρήσουν, ίσως να αλλάξουν κάποια πράγματα, λαμβάνοντας υπόψη ε, ε, κάποιες περαιτέρω ε, πλευρές. Επίσης υπάρχει μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με τις συλλογικέ συμβάσεις που κάνουν αναφορά στην προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι συμβάσεις να ληφθούν υπόψη. Ο στόχος ο δικός μας τώρα ήταν επίσης να εξασφαλίσουμε ελάχιστα επίπεδα κανόνων. Όπως σας είπα, έχω γνώση ότι η κατάσταση ποικίλει από χώρα σε χώρα αλλά τα ελάχιστα επίπεδα που προβλέπουμε εδώ κατ' εμέ ε, δημιουργεί ένα ελάχιστο πλαίσιο που μπορεί να ε, διασφαλιστεί. Έχουμε να κάνουμε την περίπτωση όπου δεν θα γίνουν δεκτά να δοθούν δεδομένα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων. Επίσης, να μην υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ακουστικού, ακουστικής παρακολούθησης και αυτό δεν είναι αποδεκτό. Όταν επίσης ένας εργαζόμενος πάει στις, στις τουαλέτες, πάει στο χώρο αλλαγής ε, ρουχισμού να προστατεύεται. Μετά έχουμε τα θέματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλα αυτά αναφέρονται εδώ πέρα. υπάρχει το δικαίωμα παρέμβασης ε, περιορισμένο όσον αφορά τον ε, εργοδότη. Επίσης κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι η αναφορά ε, του, της προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δούμε να υπάρχει προστασία και παλήθευση ότι όντω διασφαλίζονται ε, τα επίπεδα προστασίας του εργαζομένου. Έχουμε τις περιπτώσεις ε, επιχειρήσεων που ανοίγουν σε ίδια ομάδα. Όταν ε, θα γίνεται χρήση δεδομένων θα πρέπει να γίνεται αυτό με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θα πρέπει δηλαδή να καταστρατηγείται η προστασία του ενδιαφερομένου. Αυτό το βλέπουμε στο κεφάλαιο 5. Ένα άλλο θέμα το οποίο δημιουργεί πολλές ε, ε, αντιπαραθέσεις είναι ε, το θέμα το πώς α, α, τη θέση του εργαζομένου. Φερρυπίν. Έχουμε προγράμματα για άτομα που ε, ε, έχουν στην προστασία τους παιδιά. Εμείς διαβάζουμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν οικονομικές πτυχές που έχουν να κάνουν με το εργαζόμενο. Είχαμε περίπτωση συγκεκριμένου παραδείγματος. Ε, έγινε μία εξέταση με τον εργαζόμενο να παληθευτεί, φέρει πει, αν το παιδί βρίσκεται στο παιδικό σταθμό και αν ε, ε, υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα για το εργαζόμενο ή όχι. Ήταν κάποια από τα παραδείγματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορούμε φυσικά να δούμε ανάλογες περιπτώσεις και σε άλλους τομείς. Ε, επίσης, για την εκπροσώπηση. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί να τα αλλάξει τα πράγματα η Επιτροπή. Είναι πολύ λεπτά θέματα. Δεν μπορεί να παρέμβει ε, τόσο εύκολα επιτροπή. Έχουμε να κάνουμε θέματα ασφάλειας, τεχνικής ε, πτυχής και η Επιτροπή θα πρέπει με διαβούλευση να, να δημιουργήσει καινούριους, να καθορίσει καινούριους στόχους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η προστασία του ενδιαφερμένου. Αυτά σε γενικές γραμμές, στα πλαίσια πάντα του άρθρου 82, έτσι δουλέψαμε. Είναι όμως ένα θέμα αυτό για την προστασία των δεδομένων τόσο σημαντικό που πραγματικά αξίζει να το δούμε πιο ευρέως. 11 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες συμβαστικές ε, προτάσεις. Είναι δύο ισχυώδεις συγητές. Ξέρουμε πραγματικά. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος, Αλεξάνδρος Σέρκας και η κυρία Μακεντάιρ. Ζητώ συγγνώμη που είπε λάθος το όνομά σας. Αυτούς έχουμε προς το παρόν. Θα ήθελα να μιλήσει και κάποιος από την Κομισιόν στη συνέχεια, ναι. Ωραία, η Κομισιόν λοιπόν θα παρεμβεί μετά. Αλεξάνδρος Σέρκας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ο σκιώδης ε, εισηγητής μας λόγω της αλλαγής της ώρας παρουσίαση αυτού του θέματος δεν καταφέρει να βρίσκεται εδώ σήμερα. Μου άφησε λοιπόν κάποιες σημειώσεις ε, και κάποιες προφορικές οδηγίες. Ε, πρώτα απ' όλα η γνωμοδότησή μας, η, η άποψή μας είναι πολύ ευνοϊκή διότι από πολύ πρώιμο στάδιο η κυρία Χέρς ήρθε σε επαφή με τους και έγιναν σημαντικές αλλαγές και βλέπουμε στις τροπολογίες σας ότι λάβατε υπόψη όλους τους ενδιασμούς που είχαμε σε σχέση με αυτό τον εξαιρετικά σημαντικό φάκελο για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω επ' αυτού ότι εμείς επικεντρωθήκαμε σε τέσσερα σημεία, δηλαδή τη δυνατότητα των κρατών μελών να καθιερώνουν ελάχιστα επίπεδα και αυτό ερμηνεύεται πολύ ευνοϊκά. Τώρα Όσοι ασχολούνται με την προστασία των δεδομένων και είναι επιφορτισμένοι με αυτό και αυτοί πρέπει να προστατεύονται κατά οποιασδήποτε πίεση από εταιρείε ή οποιονδήποτε άλλον. Όλο αυτό το κομμάτι του ιδιωτικού απορρίτου των εργαζομένων πρέπει να προστατεύεται με την καθιέρωση αυτών των κανόνων. Πρέπει να διακρίνουμε την εργασία και την ιδιωτική ζωή. Όπως είπατε λοιπόν, οποιοδήποτε μυστική παρακολούθηση πρέπει να απαγορεύεται αυστηρά. Τώρα όσον αφορά τα στοιχεία που καλύπτουμε εδώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες ουσιαστικά το άρθρο 82 π. δεν είναι επαρκές για να προστατεύσει τόσο πολλά συμφέροντα δεδομένου του διακυβεύματος και μπορώ να σας δώσω και μια εικόνα των σημαντικών ζητημάτων που θεωρούμε εμείς. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το κατόφλι των 250 υπαλλήλων σημαίνει ότι οφείλουμε τους, το 90% των εργαζομένων χωρίς προστασία. Πρέπει να βρούμε μια λύση, διότι διαφορετικά ο κανόνας αυτός δεν θα εφαρμόζεται στο 90% των Ευρωπαίων εργαζομένων. Επιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα ω εκπρόσωποι των εργαζομένων πρέπει να δώσουν την άποψή του και να συμμετέχουν στην καθιέρωση αυτών των κανόνων διότι αυτοί είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τους χώρους εργασίας τις δυναμικές των χώρων εργασία που υπάρχουν δυσκολίε, τα ζημία που δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα πιστεύουμε ότι όλοι μιλάνε, λένε πολλά και κανείς δεν γράφει τίποτα ε, κάποια ε, λίστα μαύρη ή ανθρώπων που υποστηρίζουν την προστασία στον χώρο εργασία. Έχουμε την ευκαιρία εδώ να το δημιουργήσουμε αυτό, να το στείλουμε σε εταιρείε. Αυτή η μαύρη λίστα υπάρχει και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να θέσουμε τέλος σε αυτές τις πρακτικές οι οποίες ε, βάλλονται κατά των ελευθεριών ε, της Ένωσης διότι αυτές οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν τέτοιου είδου απειλές να διαδίδονται πάρα πολύ εύκολα χωρίς κανούς είδους περιορισμού. Και είναι σχεδόν αδύνατο να τις εξαλείψει κανείς. Ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό για μας το μελετάμε μάλιστα πολύ στενά και ξέρω και οι κυριαρχές και θα συνεχίσουμε να έχουμε υπόψη μας ότι σε περίπτωση διένεξης ή διαφωνίας, διαφοράς όσον αφορά μεταξύ επιχείρηση και εργαζομένων. Υπάρχει διένεξη όσον αφορά θεμελιώδη δικαιώματα εργαζομένων, όσον αφορά τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα. Ε, εδώ μιλάμε για ένα κανόνα προστασία και η αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά περίπλοκου ζητήματο, όλοι μα, όλε τι ομάδε και ο η εισηγήτρια θα πρέπει να συνεργαστούμε ώστε να ε, καταλήξουμε σε ένα πολύ καλύτερο κανόνα και πιστεύω ότι μπορούμε να το ε, επιτύχουμε. Κυρία Μάκεντάιρ. Um, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για τη δουλειά της αυτή, την γνωμοδότηση και για τη συνεργασία της. Ε, Ανυπομονώ να συνεργαστούμε στι συναντήσεις των σκιωδών. Πιστεύω ότι στόχος του κανονισμού είναι να παρέχει ε, σαφήνεια για τις επιχειρήσεις ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να γνωρίζουν τι απαιτείται από αυτέ. Εάν λοιπόν αυτός, ο κανονισμός πρόκειται να περιλάβει το αρθρό 82 για την απασχόληση, θα πρέπει να είμαστε σαφείς στο τι ζητάμε να κάνουν τα κράτη-μέλη να μην ε, θέτουμε υπερβολικούς όρους και κυρίως να είμαστε σαφείς προς τις επιχειρήσεις. Και πάντα το αναφέρω αυτό, οι μικρές επιχειρήσεις και οι μικροεπιχειρήσεις υποφέρουν από την έλλειψη σαφήνεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν ήδη θεσπισμένη νομοθεσία που λειτουργεί καλά για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι η πρότασή μας δεν θα περιορίσει αυτό που κάνουν ήδη τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε την ανάλογη ευελιξία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, χρειαζόμαστε υψηλό επίπεδο και πρέπει να παρέχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει σε άλλα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν επαρκή προστασία δεδομένων να δημιουργήσουν αυτή την προστασία. Θεωρώ ειδικότερα για, στο, με το άρθρο 82 εμείς ανησυχούμε που δεν αναφέρεται καθόλου η διαφάνεια, η αναλογικότητα των πληροφοριών. Δεν λέγεται τίποτα για την ασφάλεια των δεδομένων και τίποτα σε σχέση με την ευαισθητοποίηση, σε σχέση με τις πληροφορίες που υπάρχουν. Δηλαδή να γνωρίζει το προσωπικό της εκαστή εταιρείας τι πληροφορίες λαμβάνονται, διατηρούνται από την εταιρεία. Ωστόσο Κύριο μας μέλημα είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε η Κομισιόν να έχει, να έχει τη δυνατότητα κατεξοδότηση πράξης ε, στον τομέα της απασχόλησης ε, με ανεπιθύμητα αποτελέσματα ε, όπου θα μπορούσε η Κομισιόν να αλλάζει κάποια πράγματα πολύ γρήγορα. Αυτό μας ανησυχεί κυρίως. Υπάρχουν περίπου ε, πάνω από 90 κατεξοδοτήσεις πράξεις σε αυτόν τον κανονισμό, πολύ περισσότερες από την φυσιολογικό και πιστεύω είναι σημαντικό να επιτύχουμε μια καλή ισορροπία ώστε να μην υπερφορτώσουμε το κείμενο αλλά ταυτόχρονα ή, τις επιχειρήσεις ε, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλουμε απλά να δώσουμε κατεξοδότηση πράξη ελεύθερα στην Κομισιόν ανυπομονώ να συνεργαστούμε και να εξετάσουμε τις τροπολογίες που θα σας υποβάλω. Ευχαριστώ. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ. Τόμα Σέρδικ, ονομάζομαι, εκπροσωπώ την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνη και ασχολούμαι με τα θέματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, Χαιρετίζουμε την δέσμευση που του Κοινοβουλίου που διαπιστώνουμε μέσα στη γνωμοδέτηση της κυρίας Χίρς ε, για να προωθήσει αυτό το ζήτημα. Η, εν γέννη είναι αγαστή η συνεργασία μας. Τώρα ιδιαίτερος ε, για το μεταρρυθμιστικό αυτό πρόγραμμα, όπως σωστά μας είπε η συγγήτρια είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη, αλλά και για την Επιτροπή. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μισθωτών. Λοιπόν, εξετάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τις προτάσεις σας και διαπιστώνουμε πως η κυρία πραγματεύεται ε, βασικά ζητήματα προστασίας των δικαιωμάτων ε, των εργαζομένων ε, στα πλαίσια του κανονισμού. Γνωρίζουμε ότι η οδηγία 9546 είναι αυτή που διέπει το ζήτημα και ο κανονισμός ενέχει διεξοδικότερες διατάξεις για το ίδιο ζήτημα. Προβλέπεται Ε, αναβαθμισμένη, ενισχυμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν θα επιδεινωθεί η κατάσταση ως προς την προστασία των δεδομένων. Τώρα, αν τα κράτη-μέλη επιθυμούν ισχυρότερη προστασία, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και αυτό συμφωνεί και με τον δεδηλωμένο στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασιζόμαστε στην κείμενη νομοθεσία, την οδηγία 95 και σε καμία περίπτωση η οδηγία αυτή δεν πρέπει να θέσει ένα αμφιβόλιο την ελεύθερη το δικαίωμα ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Εξετάζουμε επίση ε, τι ε, συμφωνίε ε, για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει στο μέτρο που είναι πηγή δευτερογενούς ε, δικαίου. Μας απασχολεί επίσης το θέμα του ρόλου των μισθωτών μέσα στην επιχείρηση. Ήταν ένας από τους στόχους μας. Θα θέλαμε κάποιους ε, ε, επικεφαλής της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα εξασφαλίσουν ότι η χρήση των δεδομένων αποσκοπεί στην ευημερία των μισθωτών αλλά και ε, στην προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Το άρθρο 36, εδάφιο 2, και το αναφέρω επειδή αναφερθήκατε και εσείς σε αυτό το άρθρο, προβλέπει ακριβώς αυτή τη δράση. Ακολουθήσαμε την λογική αυτού του άρθρου. Για την ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών ε, μέσα σε ε, κοινοπραξίες επιχειρήσεων, ε, υπάρχουν σχετικές νομικές διατάξεις που διαφυλάττουν το δικαίωμα της επιχείρησης να μετακινεί τους μισθωτούς Πρόκειται για το άρθρο 6.1 σίγμα Συμφωνούμε με τις γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθείτε, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για τις τροπολογίες που έχετε καταθέσει. Θα ήθελα όμως να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην υπάρξουν αντιφάσεις με τις λοιπές διατάξεις του κανονισμού. Ένας άλλος στόχος είναι η δράση μας να μην οδηγήσει σε ανεπιθύμητες ε, για τους μισθωτούς ε, επιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, χρειάζεται και προβλέπεται η συγκατάθεση του μισθωτού σε κάποιες περιπτώσεις ε, δεν θέλουμε πάση θυσία να αποφύγουμε το να παρακάμπτεται η νομοθεσία. Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθω για τις τροπολογίες. Ε, ευχαριστώ. Μας ακούσουμε την εισηγήτρια μου. Ähm, ευχαριστώ για, ευχαριστώ και για τις παρατηρήσεις που κάνατε. Θα επανέλθω σε κάποια θέματα. Ο κύριος Σαρκάς έκανε κάποιες αναφορές. Υπάρχουν και άλλες πτυχές αυτού του κανονισμού που αφορούν τους εργαζόμενους. Όπως είπαμε, όπως ελέγχθη από πολλούς, θα κατατεθούν τροπολογίες. Ο στόχος μου είναι να μην ε, θα πρέπει να γίνει η δυνατότητα να ακουστούν και απόψεις της δική μας Επιτροπής στα πλαίσια του άρθρου 82 υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία κυκλοφορούν ε, και στις άλλες επιτροπές και δεν είναι σωστό να ορίσουμε ε, μια, ένα, να κάνουμε ένα περιορισμό κάποια όρια και να αποκλειστεί η πλειοψηφία. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε μια ενδεχομένω άλλη διατύπωση, λαμβάνοντα υπόψη το γενικότερο πλαίσιο και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια, την καλύτερη δηλαδή μάλλον διατύπωση. Όταν θα έχω τις τροπολογίες θα δω τι μπορώ να κάνω. Αλλά επιμένω, το 82 είναι το πιο σημαντικό άρθρο και θα πρέπει να το βάλουμε στο κέντρο όσον αφορά τις δικές μας ε, ανησυχίες. Υπάρχει φυσικά και το θέμα των μαύρων καταλόγων που δεν πρέπει να υπάρχουν, αυτό που λέμε μαύρη λίστα. Εμείς, όπως και να έχει το θέμα, εμείς θα προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο, να τα αποκλείουμε αυτά. η κυρία Μακεντάιρ έθιξε ένα άλλο πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε διαφορετικές συνθήκες από μία χώρα στην άλλη. Φυσικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουν να καταλήξουν σε ένα επίπεδο ε, που μπορεί να τους οδηγήσει σε, μια, σε περαιτέρω ας πούμε βάρος διοικητικό. Θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Θα το λάβουμε υπόψη. Όσον αφορά δε τις κατεξιοδότηση πράξης, θα πρέπει και εδώ να δούμε ποιες είναι αυτές οι πράξεις που επιθυμεί το Κοινοβούλιο και ποιες δεν θέλει, ποιες είναι κατεξιοδότηση πράξης οι πιο σωστές, οι πιο σημαντικές ούτως ώστε να μην αποκλεισούμε εντελώ από τη διαδικασία. Θα πρέπει δηλαδή να ταξινομήσουμε τις διάφορες καταξιοδότηση πράξεις. Ευχαριστώ όμω σε γενικές γραμμές όλες τι παρατηρήσεις και την Επιτροπή και στα μέτρο του δυνατού θα κοιτάξουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, την μέγιστη δυνατή λύση. Και όπως καταλάβαμε θα πρέπει να πανεξετάσουμε κάποια θέματα. Δεν μας δημιουργεί αυτό προβλήματα. Όπως είπε ο κύριος Σαρκάς, είναι να έχουμε ένα σωστό έγγραφο, ένα δυνατό άρθρο 82 για να μπορέσουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προστασία. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Τώρα, 11 Δεκεμβρίου, Τρίτη, κατάθεση τροπολογιών, προθεσμία δηλαδή. 24 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε το θέμα. 20 Φλεβάρι θα κοιτάξουμε τις τροπολογίες, μετά προσπαθήσουμε να ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Είναι, αυτό το πρωινό είναι της κυρίας Μακεντάερ, η οποία θα πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει 199 τροπολογίες που κατατέθησαν στη δική της πρωτοβουλίας όσον αφορά την ενσωμάτωση των μεταναστών, συντονισμούς σε σχέση με θέματα κοινωνικής ε, ασφάλειας. Είναι οι εκθέσει ΑΦΕΤ και γυναίκες έχουν ε, αναλάβει γνωμοδότηση επιπλέον. Έχουμε σε αυτή την έκθεση μία διαδικασία, διαδικασία σε συνεργασία με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την οποία ο διοικητής ε, για την γνωμοδότηση, ο Φίλιπ Κλέης, ε, και ο οποίος δεν ξέρω αν είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή, όχι, δεν τον βλέπω. Αυτός θα συνεργαστεί εγγράφος. Παρακαλώ να δώσουμε το λόγο στην κυρία εισηγήτρια τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις τροπολογίες. 199 ήταν οι τροπολογίες για διάφορα θέματα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η ανάγνωση όλων αυτών των τροπολογιών. Ε, εγκρίναμε όσε τροπολογίε μπορούσαμε δεδομένες τη ποικιλομορφία του. Δεν θα σα τις παρουσιάσω λεπτομερώς. Ε, απλά Ήθελα να αναφέρω κάποια προβλήματα με ορισμένε τροπολογίε που αφορούν κυρίω τι αρμοδιότητε τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τα δικαιώματα των μελών τη οικογένεια. Ε, θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να τι ενσωματώσουμε στην πρότασή μα. Ε, κατά τα άλλα, ε, η μεγάλη πλειοψηφία το... θα προσπαθήσω να ε, συμπεριλάβω σε συμβιβασμού τις περισσότερες τροπολογίες ε, διότι αφορούν παρόμοια θέματα υπάρχουν αντιθέτω, κάποιε άλλε τροπολογίε που κινούνται προς εντελώ αντιθετή κατεύθυνση πολύ πιο περιοριστικέ. θα ήθελα λοιπόν να δείξετε κατανόηση δεν μπορώ να τι λάβω υπόψη στι συμβιβαστικέ λύσει, διότι κινούνται προς εντελώ αντίθετη κατεύθυνση στη συνέχεια υπάρχουν και προβλήματα μετάφραση, διατύπωση. Όταν μιλάμε λοιπόν για πιθανά ε, πιθανές ικανότητες, πιθανά ταλέντα στα γερμανικά μερικές φορές ε, έχει μεταφραστεί πολύ λάθος θα πρέπει να βρούμε λοιπόν άλλες ερμηνείες ώστε να κατανοήσουμε καλά τι εννοούμε με αυτή τον ορισμό το ζήτημα των παράνομων μεταναστών μπορούμε να το αλλάξουμε σε regular migrants ε, ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών ε, και των ομοφιλοφίλων έγινε μια πρόταση κατάργησης δεν θα ακολουθήσουμε αυτή την πρόταση αλλά θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια παράγραφο πλήρη για αυτά τα ζητήματα στη συνέχεια είχαμε και την τροπολογία 33 η οποία αφορούσε για ethnic business. Ε, εσπίζουμε ότι καταλάβαμε καλά, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε γι' αυτό για να, να δούμε τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Είχαμε μια μεγάλη σειρά τροπολογιών για διάφορους τομείς. Εμείς θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε συμβιβαστικές τροπολογίες. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίσαμε το ζήτημα θεματικά ουσιαστικά κατά θέματα διάφορες τροπολογίες βλήθηκαν και διάφορες παραγράφους και εμείς προσπαθήσαμε να μην χειριστούμε αυτές τις τροπολογίες κατά παράγραφο αλλά κατά θέμα. Δηλαδή, η τροπολογία σα μπορεί να μην αναφέρεται στην αρχική παράγραφο στην οποία αναφερθήκατε, αλλά σε κάποιο άλλο σημείο που μα φαίνεται να αρμόζει καλύτερα. Έχουμε προβλέψει δύο ε, συνεδριάσεις σχεδόν εισηγητών την επόμενη εβδομάδα η πρώτη και στη συνέχεια θα λάβετε τις συμβαστικές τροπολογίες. Στη συνέχεια θα έχετε αρκετό χρόνο να εξετάσετε αυτά τα έγγραφα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ καλά και εξαιρετική συνεδρίαση και οδό Συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη τώρα γιατί πέφτει πάνω σας αυτό που θα πω. Εγώ προεδρεύω στις εργασίες εδώ και το έχω πει επανειλημμένα. Πρέπει να μεριμνούμε ώστε να είναι ποιοτικές συζητήσεις μας και στην Ολομέλεια. Εάν ασχολούμαστε μόνο με τυπικά και διαδικαστικά ζητήματα, τότε ε, ε, δεν θα έχουν νόημα οι συνεδριάσεις ολομέλειας επιτροπής μας. Ε, αυτό μπορεί να γίνει στι ομάδε εργασία ή στου καφέδε που πίνουμε με του συναδέλφου ε, για να καταλήξουμε σε συμβασμού. Ε, είναι και αυτά σημαντικά, αλλά ε, για την ποιότητα των εργασιών μας και για να τροφοδοτούμε τον προβληματισμό των βουλευτών με ορθό τρόπο, πιστεύω ότι πρέπει να διεξαγόνται διαφορετικά οι εργασίες. Δηλαδή, είναι ανοιχτές στο κοινό αυτές οι συνεδριάσεις και είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Τώρα εξετάζουμε τι επιπτώσει ε, τη ε, αδίλωτης μετανάστευση στην εσωτερική αγορά. Μα είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα και εφόσον είχαμε την ευκαιρία ε, να ακούσουμε την παρουσίαση και τις κατευθυντήριες γραμμές της εισηγήτριας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα στη συνέχεια των διαπραγματεύσεων. Θα συμφωνήσει και η εισηγήτρια νομίζω μαζί μου. Ε, πραγματικά νιώθω... Δεν είμαι ικανοποιημένη από αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων. Όσοι παρακολουθούν τις εργασίες μας ε, ε, στο διαδίκτυο ή μέσα στην αίθουσα, νομίζω αυτό περιμένουν ο σκιώδης εισηγητής που έχει το προνόμιο να είναι στο κλάστερ στην ομάδα των διαπραγματευτών δεν είναι δυστυχώς εδώ, αλλά έχουμε την κυρία Γιάσλοβίσκα η οποία θα τον αντικαταστήσει και η κυρία Μπλίνκεβιτσε θα πάρει ε, στη συνέχεια το λόγο. Παρακαλούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που απουσιάζει ο συνάδελφος. Δυστυχώς, αναγκάστηκε να παραμείνει στη Ρουμανία και δεν ε, μπόρεσε να έρθει για τη σημερινή συνεδρίαση. Διακόπτει ο Είναι κατεπήγον το ζήτημα της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας. Ε, με την κατάσταση που βιώνουμε τώρα συνειδητοποιούμε ότι Υπάρχει ύφεση στις οικονομίες μας ε, και για να τονώσουμε την οικονομία θα πρέπει να υιοθετήσουμε και μια ε, πιο ανοιχτή προσέγγιση για την ενσωμάτωση αυτών ε, των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιδιώκουμε μια πιο ανοιχτή αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύπτονται οι κενές θέσεις από αυτούς τους εργαζόμενους. Έχω καταθέσει σχετικές ε, τροπολογίες για να χρησιμοποιηθεί η παιδεία, η ενημέρωση ως προς τις επαγγελματικές δεξιότητες για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, να συνιστούν δηλαδή προϋποθέσεις ώστε να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να υπάρχει καλύτερη αντιστοίχηση τη προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Η επιδίωξη των καταλήλων επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη συνιστόσα αν επιθυμούμε να ενσωματώσουμε στην αγορά εργασίας μας ε, εργαζόμενους από τρίτες χώρες ε, που έχουν μετικήσει στην Ένωση. Κάτι άλλο σημαντικό, η οικονομική, η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι ήπιες αναπτυξιακές μεσοπρόθεσμες προοπτικές δημο διαμορφώνουν μια κατάσταση όπου κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις επιπτώσεις ενσωμάτωσης αυτών των ανθρώπων λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται σωστά η κείμενη νομοθεσία. Δεύτερον, οι εξελίξεις στην αγορά εργασία σε επίπεδο κρατών μελών παρουσιάζουν σημαντικότατες αποκλήσεις αυτή τη στιγμή. Και άρα θα πρέπει με στόχο πάντοτε την ενσωμάτωση αυτών των εργαζομένων να εξασφαλίσουμε προστιθέμενη αξία για τις ε, οικονομίες μας και όχι περαιτέρω προς κόμματα. Ε, μην ξεχνούμε ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν και πολιτικές επιπτώσεις. Είναι ευθύνη μας ε, να ενημερώσουμε σωστά και να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα στους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της απροθυμίας κάποιων κρατών μελών για το άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε αυτούς τους εργαζομένους, κρίνω ότι είναι κέρια σημασία μείνουμε σε αυτόν τον στενό διάλογο με τα κράτη-μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ε, για το ζήτημα αυτό, μειώνοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του είδους της μετανάστευσης. Ε, και θα ήθελα να προσθέσω ότι αν ε, ρυθμίσουμε σωστά το ζήτημα της ενσωμάτωσης τους, ε, θα ε, επωφεληθεί από αυτό και η ευρωπαϊκή οικονομία. Ξαναλέω, πρέπει να σεβόμαστε την κείμενη νομοθεσία, να έρουμε τους ε, περιτούς φραγμούς, να ανοίγουμε την αγορά εργασίας με τρόπο ώστε να είναι υποφελής η κατάσταση και για τους εργοδότες και για τους όσους ε, επιθυμούν να βρουν μια θέση απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αλλάξω τώρα γλώσσα, ε, διότι δεν μιλώ πλέον εξ ονόματος του συναδέλφου μου. Θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, το ζήτημα της ενσωμάτωσης ε, αυτών των εργαζομένων επηρεάζει ε, σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα στην αγορά εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω καταθέσει τροπολογίες, ε, των οποίων το βασικό μήνυμα είναι το εξής. Είναι κατεπήγον το να ε, πληρούνται οι κενές θέσεις στην αγορά εργασίας και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει με επιτυχία να ενσωματώσουμε υπηκούς τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας ε, της Ένωσης. Αυτό σε μια πρώτη φάση και σε μια δεύτερη φάση να ενσωματώσουμε ε, και τους εργαζόμενους που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προωθήσουμε επίσης το θέμα της αναγνώρισης ε, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Δεξιοτήτων που δεν εφαρμόζεται ικανοποιητικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιείται ήδη το σύστημα για τους υπηκούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να επεκτείνουμε την εφαρμογή του και στους υπηκούς ε, τρίτων χωρών. Επίσης, Χρειαζόμαστε ε, συστήματα με τα στοιχεία ε, αυτών των ε, εργαζομένων για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μηχανισμούς στήριξης των εργαζομένων αυτών. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλους τους ενδιαφερομένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος συγγνώμη, κυρία Μπλίντσεβούτε πήρε το λόγο απευθεία. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση της Νάντια ε, είναι πολύ δημοφιλής. Πάνω από 200 τροπολογίες υποβλήθηκαν και θα έλεγα ότι η έκθεση θα είναι καλή. Είμαστε πολύ υπέρ αυτής της έκθεσης. Δύο παρατηρήσεις. Θα ήθελα και εγώ να βρεθεί μια συμβαστική λύση ώστε να ενθαρρυνθούν οι μετανάστες επιχειρηματίες. Είναι σημαντικό μετανάστες από τρίτες χώρες όχι μόνο να δημιουργούν θέσεις εργασίας αλλά και να ενθαρρύνουμε κοινωνική κινητοποίηση και κοινωνική συνοχή. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ένα άλλο σημαντικό σημείο αφορά, όταν, αφορά, όταν μιλάμε για την ένταξη ενσωμάτωση των μεταναστών είναι η κατάρτιση των εργαζομένων των μεταναστών, η πρόσβαση σε κατάρτιση και εκπαίδευση υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν μερικές φορές σε εκπαιδευτικό επίπεδο χαμηλότερο από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά των οικογενειών μεταναστών να ακολουθούν ε, κάποια εκπαιδευτικά εκπαίδευση. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι έτοιμα να δουλέψουν με τα παιδιά των ε, μεταναστών. Ε, θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάτι στη... όσα είπε η κυρία Νάντια Χέρς όχι μόνο ε, οι χώρες ε, ε, προέλευση θα πρέπει να είναι υπεύθυνε, οι, οι, οι χώρες υποδοχής των μεταναστών πρέπει να έχουν την αρμοδιότητα ένταξης των μεταναστών παρέχοντας τους εκπαίδευση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα ενσωμάτωσης έτσι. Όταν μιλάμε για ευθύνη, για επιτυχή ένταξη πρέπει να εστιαζόμαστε στις χώρες υποδοχής. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τους συναδέλφους να εξετάσουν το ενδεχόμενο ε, προγραμμάτων διαβίου μάθησης και προγραμμάτων κινητικότητας ε, που παρέχονται σε τρίτες χώρες. Όσον αφορά το σύστημα βαθμών που προτείνει, το point system που προτείνει η συγκήτρια, το πρόβλημα εκεί είναι, κατά την άποψή μου, ότι αυτό το σύστημα δεν είναι ακόμα σαφές, δεν είναι σαφές πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα λειτουργήσει στα κρατη Έχει κάποιες ελλείψεις και δεν είμαι βέβαιη κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να προσφέρει προς τη θεμενή αξία, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση σε σχέση με αυτό το point system ίσως να μην προτείνουμε εφαρμογή του συστήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά πιστεύω ότι στη συνεδρία και εδώ είναι θα καταφέρουμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Ευχαριστώ. Jean Lambert. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πω και πάλι ότι είχαμε την εντύπωση ότι η αρχική έκθεση ήταν πολύ καλό εφαλτήριο, όμως λαμβάνοντας τις τροπολογίες διαπιστώνουμε σημεία διένεξης γύρω από τις παραγράφους 7 και 8. Έχουμε και κάποιους ενδιασμούς, όπως είπε η Μπλίνκετ Σουβίτε, για το θέμα το... της βαθμολόγησης. Μπορούμε να βρούμε μία λύση. Ίσως στην παράγραφο 29 και στην παράγραφο 28 για τα συστήματα κοινωνικής ε, ασφάλισης ε, δεν μας τρελαίνει αυτή η ιδέα, στο θέσω έτσι. Έχουμε εναλλακτικέ ε, προτάσει. Υπάρχουν και κάποιε σκληροπυρηνικέ τροπολογίε για τη διαγραφή του σημείου, αλλά πιστεύω ότι οι σκιώδει θα καταφέρουν να βρουν μια λύση. Καταθέσαμε τροπολογίες λοιπόν για τη διάσταση της κοινωνικής ασφάλισης ε, για αυτή την έκθεση. Ε, στην ε, τροπολογία 182 και εξής αυτοί οι κυκλοφορούντες μετανάστες, έτσι τους ονομάζουμε και αυτοί ε, που διέρχονται τα σύνορα κρατών της Ένωσης αλλά παραμένουν στο εσωτερικό της Ένωσης λοιπόν μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια σειρά διμερών συμφωνιών με τις χώρες προέλευσης κυρίως θα μιλάμε για κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τρίτες χώρες υπάρχουν ε, ε, μόνο οι διμερείς συμφωνίες σε επίπεδο κρατών μελών ως προς τη συνεργασία των εμπειρογνωμών των κρατών μελών ε, που ασχολούνται με αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Πιστεύω αυτή θα ήταν μια καλή ιδέα για να σχεδιάσουμε τις μελλοντικέ μας κινήσεις. Επίσης, ε, άρση φραγμών σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών ε, για λόγους που σχετίζονται με την ξενοφοβία και το ρατσισμό. Οι προτάσεις που κάναμε έχουν ήδη ενσωματωθεί. Διάφορες τροπολογίες όπως και άλλοι κατατέθηκαν για το ρόλο των εργοδοτών για την ενσωμάτωση των μεταναστών, μιλάμε για την αγορά εργασίας και ε, ως εκ τούτου πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ε, τι ποια συνιστά ευθύνη των εργοδοτών και τι συνιστά ευθύνη άλλων. Άρθρο 62, ρόλος άλλων φορέων για ε, το θέμα της ενσωμάτωσης, ε, πρόσβαση στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Ξέρω ότι ε, συζητήθηκε το θέμα με τα κράτη-μέλη και σε σχέση με άλλες προτάσεις και με ξαφνιάζει που όλοι επιθυμούν οι μετανάστες να μάθουν τη γλώσσα της χώρας αλλά δεν υπάρχουν τόσα διαθέσιμα μαθήματα. Η αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων πιστεύω είχε αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και τις τροπολογίες 1, 2, 3 που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Ε, είμαι σίγουρη ότι σε συνεργασία με τους υπολείπους ε, θα καταλήξουμε συμβαστικές ε, λύσεις η πρόταση της ε, εισηγήτριας, ε, δηλαδή να ε, υιοθετήσουμε θεματική προσέγγιση για τις τροπολογίες, αντί να τις εξετάζουμε κατά περίπτωση, όπως συνέβαινε στην αρχική σας έκθεση, Νάντια, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, διότι έχουμε τελίτσες και σταυρουδάκια παντού και πρέπει να θεματοποιήσουμε, να ομαδοποιήσουμε τις τροπολογίες σας. ευχαριστούμε πάντως για την καλή συνεργασία και προσβλέπουμε στην μελλοντική ε, συνεργασία που θα μας οδηγήσει, ελπίζουμε, σε μια επιτυχημένη γνωμοδότηση και ε, όσοι επιθυμούν μπορούν να δουν και τι συμβαίνει στην Επιτροπή Προσωπικών Ελευθεριών. Πρόεδρος, ε, υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο, παρακαλώ, για αυτό το θέμα. θα ξανακούσουμε την εισηγητριά μας, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις τόσο διαφορετικές ε, παρατηρήσεις. Κυρία Πρόεδρε, ειλικρινά δεν έχω ε, δυσκολίες. Θα μπορούσα να μιλήσω για ώρα εδώ πέρα για την έκθεσή μου. Εδώ έχουμε να κάνουμε θέματα οργάνωσης. Ε, ήδη χθε το αναβάλαμε από την ημερήσια διάταξη. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα είμαι σύντομη. Είμαι όμως έτοιμη να απαντήσω στις διάφορες παρατηρήσεις. Φυσικά, για το θέμα της πρόσβασης στη γλώσσα και διαθεσιμότητα ε, κύκλων μαθημάτων. Αυτό είναι θεμελιώδες και η οποία φυσικά πολιτική ποικίλει από χώρα σε χώρα. Είναι θεμελιώδες θέμα. Αυτό θα επανέλθουμε δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με κάποιες διεκδικήσεις ότι οι μετανάστες πρέπει να μάθουν τη χώρα στην οποία καταλήγουν, αλλά ε, υπάρχουν δυσκολίες και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Ένα άλλο θέμα, η κατάρτιση, η πρόσβαση μάλλον στην κατάρτιση για τους νέους και δι για τα παιδιά. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και ξανάρχεται. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει πρόσβαση, είναι και παλιό και αυτό το επιχείρημα, και πρόσβαση στα σχολεία για να μπορέσουν να αποκτήσουν ε, περαιτέρω προσόντα συμπληρωματικά. Έχουμε να κάνουμε παιδιά τα οποία είναι από οικογένειες μεταναστών και να καταλήξουν σε υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευση. Θα πρέπει να τα βοηθήσουμε. Επίσης, ε, εθίχθη το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης μέσω συμβάσεων διμερών και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που ε, χρειάζεται εναρμόνιση. Υπάρχουν χώρες που έχουν σωστές πρακτικές, που δημιουργούν, δημιουργούν όμως παρόλα αυτά κάποιες δυσκολίες. Θα πρέπει να τις ε, αντιμετωπίσουμε. Μετά η κυκλοφορία θα λέγαμε των μεταναστών. Ε, θα πρέπει να, υπάρχουν να υπάρχει πληροφόρηση, καταλήγουν κάποιοι σε μια χώρα θα πρέπει να ξέρουμε ε, ότι θα ήταν καλύτερο κάποιοι που έρχονται από κάποια άλλη χώρα να είναι ενημερωμένοι. Ε, θα πρέπει να έχουμε πληροφόρηση, να ξέρουμε την καταλληλότητα του προ συγκεκριμένου προσώπου. Ε, υπάρχουν διοικητικές διαδικασίες που μπορούν να γίνουν ήδη από τη χώρα καταγωγής. Ένα άλλο σημείο είναι η παράγραφοι 7 και 8 όπου Άκουσα διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε δεν θα θέλαμε ακριβώ έτσι τα πράγματα, θέλουμε αλλαγέ. Είναι και εδώ. Είναι κάτι που θα το δούμε με τη συνάντηση ε, που θα γίνει με τους ισχυώδεις ηγητές. Επίσης παρατήρηση συναδέλφου για τη δημιουργία ενός πλαισίου ε, για τα προσόντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Θα μπορούσε να αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχει αυτό το λεγόμενο point system, όπως στη Μεγάλη Βρετανία. Ε, και τους πόρους που θα παραπλεύουν κανείς, ίσως ε, θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Ε, αλλά την επόμενη φορά θα είμαι πιο αναλυτική στην Επιτροπή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κλείνει προς την το θέμα. Θα συνεχίσουν ε, τις συζητήσεις 23 Ιανουαρίου προθεσμία 24 στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην ομιλία για Μάρτιο ή Απρίλιο. Ε, για μια τελευταία έτσι, επίθεση έκθεσης πρωτοβουλίας. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία. 17 και 18 είναι τα δύο θέματα είναι εδώ. Υπάρχουν εδώ οι συνάδελφοι, δεν θέλω να τους απαλλάξω, αλλά να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε ορίσει. Α. Λοιπόν, ξεκινάμε. με την έκθεση της κυρίας Μακεντάερ για την πρόσβαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση. Είναι γνωμοδότηση, υπενθυμίζω. Για την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή. Παρακαλώ, συνάδελφε, να πάλι το λόγο, κύριε Σωρή. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση. Δεν ήμουν χθε παρόν, δεν πήρα το λόγο, δεν διαμαρτυρήθηκα. Ξέρετε, όταν αλλάζει κανείς την ε, ημερήσια διάταξη, ε, δημιουργεί σύγχυση Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν ήρθαν και παρόλα που έχουμε αυτές τις αλλαγές η ψηφοφορία αρχίζει με 20 λεπτά άρα μειώνεται πάλι ο, χώρος, χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για αυτούς οι οποίοι θα περάσουν τα θέματα μετά την ψηφοφορία κοιτάξτε να μην αλλάζει η ημερησία της διάταξης θα πρέπει δηλαδή όταν ορίζεται να γίνεται σε η ημερησία διάταξη Συν, πρόεδρος είμαι πολύ ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα και είναι μια πρακτική την οποία ε, προσπάθησα να τηρήσω και δεν, ήταν, ε, δεν, ε, δεν ίσχυε με τους προκατόχους μου. Να πω ότι χθε αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί, αλλά όλοι ενημερωθήκανε, ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πάνω σε αυτό το θέμα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι με τη συνηθισμένη ας πούμε, πρακτική σε όλε τι επιτροπές ενημερώνονται τα μέλη ή οι βοηθοί του για τις αλλαγές που γίνονται στην μερίσια διάταξη. Τέλος, μια άλλη παρατήρηση τώρα για την αρχική μερίσια διάταξη. Είχε ήδη προβλεφθεί ότι το θέμα της ψηφοφορίας θα γίνει στις 10 και Όντω αλλάξαμε τη μερσία διάταξη, Χωρί όμως να αλλάξουμε ε, αυτό το θέμα. Και για το θέμα της κυρίας Χίρς ε, θα ψηφίζαμε για τις 10. Θα έπρεπε η ΔΕΜΗ να σταματήσω τι εργασίες μας για να τηρήσω αυτό το χρονοδιόγραμμα για την ψηφοφορία. Δεν παρατείνουμε αυτό το θέμα για να μην ξα... ξεπεράσουμε ακόμα περισσότερο την... το χρονοδιάγραμμα. Οι συνάδελφοι ήδη έχουν ενημερωθεί για το ότι ε, ε, για την καθυστέρηση αυτήν και προτείνω λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία μετά από αυτές τις ευκρινήσεις. Παράγραφος 1, τροπολογία νούμερο 1 της κυρία Τσούμπερ. Η συγγήτρια είναι κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο τροπολογία 2. Της κυρίας Κριντβλέσκα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 1, πάλι τροπολογία παριθμών 3 του Πολ Μέρφυ, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Στο ίδιο σημείο πάντοτε. Τροπολογία 4 της κυρίας Κριτλεύσκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συνέχεια παράγραφος διδίας υπέρ κατά αποχές δεν είναι ξεκάθαρο. Υπέρ ξανά πάλι για την ίδια τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνέχεια 2β τροπολογία 6 της ιδίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 η, η τροπολογία 4 λέει υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται συμβαστική α λέει τώρα η πρόεδρος παράγραφος 3 συμβαστική β τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 3, τροπολογία 12 του κυρίου Πολ Μέρφη. Είναι κατά η κυρία Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Εντάξει. Επαλήθευση εγώ όμως δεν έχω συνήθως την κάρτα μου για να ψηφίσω ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι οι υπόλοιποι μήπως την κάρτα σας. Θέλει κάποιος... Α, έχετε. Ένα λεπτάκι θα σας περιμένουμε τότε. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. 17 ψήφοι προς 21 κατά. Όντως απερίφθη. Λοιπόν, ε, η 13 καταπίπτει ως εκ τούτου. Ε, παράγραφος 4. Συμβαστική ΣΥ 4 πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά απόχέ. Εγκρίνεται. Και τώρα φτάνουμε στην τροπολογία 19 του Φιλιππουλών υπέρ. Κατά αποχές Εγκρίνεται. Παράγραφος 5, τροπολογία 20 της κυρίας Γιασλοβιέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μετά, τροπολογία 21, Πολ Μέρφυ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ξεκάθαρα περίφθη. Παράγραφος 5. Η τροπολογία 22 της κυρίας Μόγαν Σάχτιε με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας ε, που έγκυται στη διαγραφή του όρου legal. Υπάρχουν ενστάσεις για την προφορική τροπολογία? Όχι. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε την 22 του τροποποιηθήσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά τροπολογία 24 της Αντιπροέδρου Ινέ Τσούμπερ υπέρ. Οπ, ξέχασα και μία την κυρία, του κυρίου Ποπάκη, την τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται 24 τώρα της ε, κυρία Τσούμπερ υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Μετά Τροπολογία 25 της κυρίας ε, Σιλβάνα Ράπτη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 της κυρίας Ελιζαπέτ Μογάν Σαχτιέ υπέρ, κατά, α... ναι, ξεκαθαρό υπέρ, πάλι για την ίδια τροπολογία. Κατά. Αποχές. Ε, επαλήθευση παρακαλώ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 17 προς 21. Ε, όχι, 22. 21 ψήφι κατά. Λοιπόν, αν απορρίπτεται. 27 της κυρίας Δράπτη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 28 της κυρίας Μόγαν Σαχτιέ υπέρ. Κατά. Απόχες. Επαλήθευση παρακαλώ για την 28. Άρχεται. Πέρας. 20 προς 14 ε, και 3 αποχές εγκρίνεται. 29 ε, της κυρίας Δράπτη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6, 30 της κυρίας Τσούμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 Φιλμπενιον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά 32 του ιδίου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά, 33, η κυρία Τσούμπερ ζητάει κατά τμήματα ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου χωρίς το and other production factors, υπέρ, για το πρώτο τμήμα, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα κατά. Πίπτη και φτάνουμε στην παράγραφο 7, τροπολογία 34 του κυρίου Μπένιον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 είναι γλωσσικού χαρακτήρα, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί και φτάνουμε στην παράγραφο 7, συμβαστική δέλτα τεσσάρων πολιτικών ομάδων υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται μετά τροπολογία 39 του κυρίου Πουπάκη με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας ε, ε, διαγράφουμε το tax, την λέξη tax. Υπάρχουν ενστάσεις παρακαλώ για την προφορική τροπολογία. Δεν βλέπω τίποτα. Ψηφίζουμε για 39. Ότου τροποποιηθήσα υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται μετά ε, τροπολογία 40. Με τους ιδίους όρους, παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συμβαστική ε4 ομάδων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά, παράγραφος 8, τροπολογία 43, μπένιον υπέρ, κατά, επαλήθευση σας παρακαλώ για τροπολογία 43, άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρας. 22 υπέρ 15 κατά ξεκάθαρα εγκρίνεται και φτάνουμε. όπ είναι γλωσσικό χαρακτήρα η 44, δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Το σύνολο του κειμένου με ηλεκτρονική ψηφοφορία, παρακαλώ. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι πέρας. 35 υπέρ, 0 ψήφι κατά και 2 ε, αποχές. Συγχαρητήρια ε, στην κυρία που πέρασε και τις πέντε συμβαστικές τροπολογίες, τα κατάφερα. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό το σημείο τώρα και ε, καρκινοβατούμε επιστρέφοντας στο 17. Θα δώσουμε το λόγο και πάλι στην κυρία Μάκεντάρ για να μας ε, παρουσιάσει το νέο σχέδιο γνωμοδότησης της ε, με αποδέκτη την Επιτροπή Περιβάλλοντος στην καθήλυνα αρμόδιο που εισηγητής είναι ο κύριος ε, Τόμας Ούλιερ από το ΕΛΚ και Πρόκειται για μια πρόταση οδηγίας για τους κανόνες, βασικούς κανόνες ασφαλείας για την υγειονομική προστασία από του κινδύνους που προκύπτουν από την έκθεση σε ιονίζουσες ακτινοβολίες. Είμαστε στη διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών για αυτή την έκθεση και δυνάμει του άρθρου 31 της Συνθήκης Ευρατόμ προτού διαβιβάσει την ε, πρότασή της στο Συμβούλιο που είναι από το Σεπτέμβριο του 2011 ζητά την γνωμοδότηση της ΕΟ που απεφάνθησε 22 Φεβρουαρίου του 2012 και η τελική ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανεκρίθη στις 30 ε, Μαΐου του 2012. Θα δώσω το λόγο τώρα στην εισηγήτρια για την παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησής της που συνοδεύεται από 12 τροπολογίες προς το παρόν, εκ των οποίων 4 για το πεδίο αποκλειστικής αρμοδιότητας ε, της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχετε το λόγο, κυρία Σχέτρια, παρακαλώ. Thank you very much, Madam President. <clears throat> Um, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η εκτίση σε ακτινοβολία ε, μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Ζητώ συγγνώμη. Όπως έλεγα, όλοι γνωρίζουμε ότι η εκθέση σε ιονίζουσα ακτινοβολία ενδέχεται να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και επιζήμη για την υγεία. Υπάρχουν νόμοι που διέπουν τις ραδιενεργές ουσίες και προστατεύουν τους εργαζόμενους από το 1959. Το σχεδίο οδηγίας επιδιώκει να απλοποιήσει τις υπάρξεις διευθετήσεις και συγκεντρώνει τις διάφορες οδηγίες. Νομίζω ότι υπάρχουν πέντε οδηγίες τη συγχωνεύει σε μία. Επίσης ε, συμπεριλαμβάνει τα φυσικά ραδιενεργά υλικά που είναι εξίσου επικίνδυνα με τα υπόλοιπα. Γενικά υποστηρίζω την πρόταση, τις προτάσεις της Κομισιόν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια προσέγγιση βασισμένη στην επικινδυνότητα και σε αποδεκτικά στοιχεία και να λαμβάνουμε υπόψη τις ε, πιο πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες. Γνωρίζω από συζητήσεις που έχω ήδη κάνει ότι πάντα εμφανίζονται νέα κείμενα. Νομίζω εν μέρη από την ε, ICRP που είναι η Διεθνής Επιτροπή Ακτινοπροστασίας. Προστασίας και πιστεύω ότι αναμένουμε ένα άλλο κείμενο ακόμα πριν το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας. Η γνωμοδότησή μας μπορεί να βασιστεί μόνο στην πρόταση του Σεπτεμβρίου 2011. Σκοπεύω όμως να μελετήσω τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες πριν λήξει η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Και όπου αυτό είναι δυνατό θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω τους τελευταίους προβληματισμούς ε, στις τροπολογίες, ε, στο σχέδιο γνωμοδότησής μου. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν εξαιρετικά περιορισμένο. Ο χρόνος μεταξύ του σημείου όπου η Επιτροπή μας λαμβάνει γνώση για ποια άρθρα έχει αποκλειστική μερική ή καθόλου αρμοδιότητα και ο χρόνος μεταξύ αυτού και της προθεσμίας εκπόνησης της ε, γνωμοδότησης ήταν πολύ σύντομος και αποτελεί μεγάλη πρόκληση το να εκπονήσει κανεί μια καλή γνωμοδότηση. Τώρα δεδομένων αυτών η Επιτροπή ΕΜΒΗ παράτηνε το χρονοδιάγραμμά της. Έχοντας αυτό υπόψη, δεν χρειαζόταν λοιπόν να βιαστούμε. Εμείς τηρήσαμε την προθεσμία, αλλά αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι τώρα η 10η Ιανουαρίου. Όχι μόνο λοιπόν ελπίζω ότι όλοι οι σκιώδεις θα συμμετέχουν με τις τροπολογίες τους και εγώ θα υποβάλω τροπολογίες στο δικό μου σχέδιο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σάρκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της, ε, το ότι μας άκουσε, δίνει προσοχή για τα θέματα αυτά που μας απασχολούν. Το άρθρο 4 που αφορά τους ε, μαθητευόμενους, τους ασκούμενους και τους φοιτητές. Είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουμε. Παρόλα αυτά έχουμε κάποιες δυσκολίες με αυτή τη γνωμοδότηση, διότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν, έχουν, ε, δεν είναι ξεκάθαρα. Φέρει πίν τον αποκλεισμό ή την κατάργηση κάποιων πραγμάτων, τα οποία είναι ε, πολύ σημαντικά, αποφασιστική σημασία. Επί της ουσίας, θα πρέπει να έχουμε ε, διατάξεις, κανόνες ε, ελάχιστου επίπεδου για τους εργαζομένους και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι γιατί κοστίζει απλώς. Όταν μιλάμε δηλαδή για το καθαρά οικονομικά, για άτομα, κάτι που αφορά για την υγεία των ατόμων, πραγματικά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αποδεκτό. Το κόστος της κοινωνίας Φερρυπίν, όταν έχουν να κάνουμε με ατυχήματα στον χώρο εργασία, αποδεικνύεται πάρα πολύ πιο υψηλό. Θα πρέπει δηλαδή να λειτουργήσουμε προληπτικά. Ότε λοιπόν η συγγήτρια λέει ότι κάτι είναι ε, δαπανηρό, είναι κάτι το οποίο πραγματικά με φαίνει με, για το οποίο διαφωνώ. υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες τείνουν να καταργήσουν κάποιες δηλαδή υποχρεώσεις οι οποίοι, για το το λόγο ότι είναι δαπανηρές. Υπάρχει μετά ένα κίνδυνο για το να υπάρχει μια απόκληση που ακριβώς θα γίνουν σεβαστές κάποιες διατάξεις και που όχι. Έχουμε να κάνουμε την υγεία και το πεδίο εφαρμογής αυτού του κειμένου. Κυρία Εισηγήτρια, εγώ θεωρώ ότι θα μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία σε, αυτό, σε αυτή την έκθεση. Οι σοσιαλιστές όμως δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν κάποια πράγματα τα οποία μας οδηγούν στο να πάμε προς τα πίσω σε σχέση με τη σημερινό επίπεδο όσον αφορά την ασφάλεια και την ε, υγεία. Ο κύριος Μπάνιον, παρακαλώ να ευχαριστώ. Η δουλειά έγινε λίγο υπερβολικά γρήγορα μέχρι να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε για όλη αυτή την έκθεση. Το πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν γνωρίζαμε για ελλείψεις στην προηγούμενη νομοθεσία. Καταλαβαίνουμε όμως ότι τα πάντα πρέπει να αναθεωρούνται κατά διαστήματα ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ε, καλύπτουν τις τρέψεις ανάγκες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εξαιρετικό ιστορικό όσον αφορά την ασφάλεια από εμείς ακτινοβολείο. Το γνωρίζω διότι η γυναίκα μου δουλεύει ως ακτινολόγος και ξέρω ακριβώς τι περνάει σε περιπτώσεις συμβάντων, έκθεσης, ακόμα και για, σε ελάχιστες ποσότητες ή σε περίπτωση επανάληψης μιας διαδικασίας. Όλα αυτά καταγράφονται και τα πλαίσια είναι πολύ στενά. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι κατά πόσο τα νούμερα στα παραρτήματα είναι σωστά. Θα προσπαθήσω να λάβω επαγγελματικέ σύμβουλε σε αυτά πριν υποβάλω του τροπολογίε μου, διότι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε και δεν διαφωνώ με τον κύριο Σέρκα, δεν μπορούμε να κοιτάμε το κόστος αλλά αν δεν το κοιτάμε καθόλου, διαφωνώ με τον κύριο Σέρκα, ε, μπορεί να καταλήξουμε σε μια περίπτωση όπου ε, ακτινολόγοι θα δουλεύουν μια φορά την εβδομάδα. Πρέπει να είμαστε λογικοί και να υπολογίζουμε τον πραγματικό κίνδυνο παρά να λέμε απλά να είμαστε απόλυτοι στο ζήτημα κόστους και ωφελών δεν έχει λογική και δεν έχει και πρακτική εφαρμογή θα καταλήξουμε χωρίς καμία υπηρεσία υγείας στο τέλος να ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλήξουμε σε αξιόπιστα νούμερα και αξιόπιστα μέτρα ασφαλείας ε, που θα βασιστούν στο υπάρχον πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ε, Ογκουστίν Νάνσον. Ευχαριστώ το όνομά μου είναι ο Γκεστέν Λάνσος, είμαι μέλος της Μονάδας Ακτινοπροστασίας της ε, Γενικής Διεθνής Ενέργειας που είναι αρμόδια για αυτό το έγγραφο. Ήθελα να δηλώσω ότι η Κομισιόν πιστεύει πως η πρότασή τη επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ευελιξία αφενό για τα κράτη-μέλη και αναλογικότητα των απαιτήσεων σε αυτήν την οδηγία και αφετέρου με το γεγονός ότι όπως προβλέπεται από τη συνθήκη Ευρατών τα πρότυπα αυτά από το 1959 προβλέπουν ομοιόμορφη εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν δεν έχει κάποιο πρόβλημα με τις άλλες τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής εκτός από το γεγονός, η εκτός από το γεγονός ότι το νέο όριο που προτείνεται στην οδηγία που μειώνεται σημαντικά βασίζεται σε συστάσεις της Διεθνής Επιτροπής Ακτινοπροστασίας και σε αδειάσεις στα επιστημονικά στοιχεία. Αυτό αφορά τις τροπολογίες 6 και 7. Και μιλάμε για το ραδόνιο σε αυτήν την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Μακεντάερ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια που έγιναν. Εγώ θέλω να δω τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία και λαμβάνω υπόψη τα όσα είπε η Κομισιόν, λαμβάνω επίσης υπόψη την άποψη του Φιλμπένιαν ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία. Εφόσον υπάρχουν στοιχεία θα τα υποστηρίξουμε. Θα το κάνουμε μεγάλη ευχαρίστηση. Συμφωνώ απόλυτα. Χρειαζόμαστε μια ρεαλιστική, πρακτική προσέγγιση. Ευχαριστώ τον κύριο Σέρκας που με υποστηρίζει για τους εκπαιδευόμενους και τους ασκούμενους και θα ήθελα να σας καθησυχάσω. Κατά κανένα τρόπο δεν προσπαθώ να μειώσω την προστασία των εργαζομένων. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να εξασφαλίσω ότι δεν θα κάνουμε ανθρώπου να ξοδεύουν χρήματα χωρίς κανένα όφελο. Για παράδειγμα, εξετάζω το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για κεντρική βάση δεδομένων όσον αφορά τα όρια ατομικών δόσεων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα ημερολόγιο για κάθε άτομο το οποίο να γνωρίζει όπου πηγαίνει τι δόσεις έχει λάβει το να υπάρχει μια κεντρική βάση δεδομένων δεν βοηθάει τα επιμέρους άτομα. Αυτού του είδους τις ανησυχίες έχω ότι αν υπάρχει μια κεντρική βάση δεδομένων η οποία θα κοστίσει αρκετά χωρίς να έχει σημασία ποιος θα πληρώσει αυτά τα κόστη το θέμα είναι ότι δεν προστατεύεται ο εργαζόμενος πραγματικά. Αυτά είναι τα σημεία, αυτά είναι τα κόστη τα οποία θέλω εγώ να εξαλείψουμε. Αλλά αν είστε βέβαιος κύριε Σέρκας, ε, κάνω ό,τι μπορώ για να ε, προστατέψουμε αποτελεσματικά τους εργαζόμενους σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μακεντάιρ. Τώρα θα σας ανακοινώσω το χρονοδιάγραμμα. 10 Ιανουαρίου είναι η προθεσμία υποβολή τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι και 20 Φεβρουαρίου θα εξεταστούν οι τροπολογίε και οι συμβουλευτικέ τροπολογίε επίσης 20 με 21 Μαρτίου και η υιοθέτηση στην Επιτροπή Απασχόλησης το Μάρτιο επίσης. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 5 της αρχικής ημερησία διάταξης αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Μογανσάχτια. Έχετε το λόγο. Merci, Madame la Présidente. Je... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το θέμα έπρεπε να το έχουμε εξετάσει εδώ και 15 λεπτά. Ελπίζω να υπολείπεται χρόνος για συζήτηση, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το θέμα και αγγίζει άμεσα την υγεία των εργαζομένων. Πιστεύω ότι στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και να παραμελήσουμε μια συζήτηση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και που σχετίζεται με την έκθεση ε, την οποία έχω αναλάβει για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ο στόχο είναι να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων και το ζήτημα που τίθεται, θέλω να σα το υπενθυμίσω, είναι η αναδιατύπωση της οδηγίας του 2004 για την ε, υγεία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σας υπενθυμίζω ότι η οδηγία του 2004, ε, ακόμη και αν είχε εφαρμοστεί, δεν προβλέπει εξέταση MRI το οποίο είναι επιζήμιο για την υγεία των εργαζομένων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ένα δεύτερο σημείο. Ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο για αυτό το σημείο ακολούθησαν το Κοινοβουλίο, δηλαδή έχουν δώσει ως προθεσμία την 31η ε, Οκτωβρίου 2013 για να εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη. Η οδηγία μεταγραφής έχει οριστεί την για το 2013 και καταλαβαίνετε πόσο επίγον ε, είναι το ζήτημα. Ε, ήταν δυσχερής οι διαπραγματεύσεις ε, αφενός ε, διότι το Συμβούλιο διέλυσε το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εξέτασή του και οι εκπεριτροπής ε, προεδρίες ε, ήγεραν το ζήτημα της προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από διαφορετικές οπτικές γωνίες και έπρεπε να επιφέρουμε μια νέα ισορροπία στην ανάλυση του κειμένου και να σωματώσουμε αυτό το πρόβλημα των εκπεριτροπής ε, προεδριών. Χρειαστήκαμε χρόνο διότι στην αρχή ήταν αποκλίνω να αποκλίνουν σε οι θέσει των πολιτικών ομάδων, χρειάστηκε λοιπόν και να τις εναρμονίσουμε. Είχαν κατατεθεί πολλοί άριθμες τροπολογίες, 233 το αριθμό στην αρχή, στη συνέχεια 16 επιπρόσθετες όταν ανακοινώσαμε την προθεσμία υποβολής τροπολογιών και χάρη στην δουλειά των σκιωδών εισηγητών και παρεπιπτόντως τους ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ράπτη για τους σοσιαλιστές, ε, την κυρία Χάρκιν ε, από τους ε, φιλελεύθερους, Καρίν Μαντελή για τους πράσινους, και την κυρία Ανθέα Μάκινταερ για τους συντηρητικούς και τον κύριο Τούσα για την ΓΚΟΕ. Τους ευχαριστώ εγκάρδια και καταφέραμε να καταλήξουμε σε 27 συμβιβαστικές τροπολογίες. Ε, συγγνώμη, 24 συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ε, είναι Ηράκλειο το έργο. Θα σας τις παρουσιάσω λοιπόν. προέκυψαν, ε, ξαναλέω, από την ομάδα εργασίας ε, για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και από, την, ε, ακρο, από τα σχόλια του καθηγητή Ζοκολά καθώς και μία εργασία επιτόπου στο νοσοκομείο του Στρασβούργου στο τμήμα μαγνητικών τομογραφιών. και ήθελα περιπτώσεις, να απευθύνω και σε αυτούς τις ευχαριστίες μου. Αυτά έγιναν την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Θα ήθελα, ε, πρωτού περάσουμε στην ανάλυση των συμβαστικών ε, τροπολογιών, να σας πω τα δεδομένα ECNIRP ε, υιοθετήθηκαν διότι μας επιτρέπουν μία διαρκή επικαιροποίηση των δεδομένων επιτρέποντάς μας να ε, εδραζόμεθα σε ένα διεθνές γενικώς αποδεκτό πλαίσιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Είναι ένα σημείο αναφοράς που θα μας χρησιμεύσει σε διεθνή κλίμακα. Λοιπόν, συμβαστική Α. Για να αποφύγουμε την πενταετή αναθεώρηση, η οδηγία βασίζεται ε, αποκλειστικά και μόνο σε τωρινά επιστημονικά τεκμήρια. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εκ τούτου να συνεχίσει τις επιστημονικές μελέτες και την καλό να καταθέσει νέα πρόταση οδηγίας για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των ε, ιονίζων ακτινοβολιών ε, με το που θα καταστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα επιστημονικά στοιχεία υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στους σκιώδεις εισηγητές εκτός από την επιφύλαξη για τον όρο Biophysics μέσα στην ε, συμβαστική ε, Α και θα ζητήσω από την Καρίν Μαντελή που εισήγαγε αυτόν τον όρο να σχολιάσει το επίθετο αυτό biophysical effects από πλευράς των πρασίνων. Συμβαστική α, β. Θέλουμε να ε, ε, αποφύγουμε οποιαδήποτε επιδείνωση ως προς την ε, τωρινή κατάσταση για την προστασία της υγείας των εργαζομένων. Θέλουμε να διατηρήσουμε το must και οι συνυπογράφοντες έχουν συμφωνήσεις και όλες συζητητές ενώ από πλευράς όλων των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων συμβιβαστική γάμα είναι το προσφορότερο κείμενο για να καλύψουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό περιπτώσεων έκθεσης βάση της ε, πρότασης ε, Ντέλη από τους ε, πράσινους και πάλι εδώ έχουμε την συγκατάθεση των υπολείπων πέντε πολιτικών ομάδων. Συμβαστική Δέλτα πρόκειται για νέα τροπολογία, νέα συμβαστική τροπολογία με μια γλωσσική διόρθωση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαριάν Χάρκιν ε, που ε, επέφερε αυτή την διόρθωση και συμφωνούν οι υπόλοιπες πέντε πολιτικές ομάδες, δεν αλλάζουν, οι ίδιες είναι όπως και στις προηγούμενες. Ε, συμβαστική ε, τα πρότυπα Κνίρπ, όπω σας έλεγα και προηγουμένως, προς ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, διότι πρέπει να επιδιώκουμε την παγκοσμιοποίηση των ε, όρων εφαρμογής, ε, το ΕΛΚ, οι σοσιαλιστές, ε, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι έχουν να δώσει τη συγκατάθεσή τους. Συμβαστική F. Πρόκειται για τον μετρήσιμο αριθμό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τέσσερις συνυπογράφονται σκιώδεις ε, εισηγητές, διορθώνει ο Μιλήτρια, οι πέντε σκιώδεις εισηγητές έδωσαν την συγκατάθεσή τους. Ε, συμβαστική G είναι νέα αυτή η συμβαστική και ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη διαδικασία της συναπόφασης και πάλι εδώ συνυπογράφουν οι πέντε σκιώδεις. Le compromis H concerne les... Συμβαστική H, πίνακας αντιστοίχησης, ε, ούτως ώστε να γνωρίζουμε επακριβώς με ποιο τρόπο θα γίνει η μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Πάλι οι πέντε ίδιες ε, πολιτικός, ε, πολιτικές ομάδες υποστηρίζουν αυτή τη συμβαστική. Συμβαστική I, απόκληση σε σχέση με τους ιδίους στόχου. επιτρέπεται βάσει αυτής ε, της ε, συμβαστικής εξέταση με, ηλεκτρι... Ε, με τομογράφο. Το ΕΛΚ, οι φιλελεύθεροι, οι πράσινοι και οι συντηρητικοί υποστηρίζουν αυτή τη συμβαστική. Περνάω στην J. Πρόκειται για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις με το που καταστούν διαθέσιμα τα απαιτούμενα επιστημονικά στοιχεία, αποδείξεις. Θα γίνει αυτό, αλλά προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα. Προς το παρόν τέσσερι πολιτικές ομάδες έχουν δώσει τη συγκατάθεση, ΕΛΚΑ, Φιλελεύθερη Πράσινη και Συντηρητική. Συμβαστικές KLM ε, για να λάβουμε υπόψη τις ε, πληροφορίες που μας έδωσε ο καθηγητής Ζοκολά ε, μετά από την ακρόαση που έγινε για, την προσφορο... για το αν είναι πρόσφορα ή όχι τα πρότυπα ή ΚΝΙΡΠ ε, και εάν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους ε, βιοφυσικούς παράγοντες ε, στον υπολογισμό Ο κύριο Ντέλη επενεύει για αυτό το σημείο, θα μα τα πει μετά. Ε, συμβαστική εν Βασίζεται σε 30 ε, περίπου τροπολογίες ε, αυτή η συμβαστική τροπολογία και καλύπτει τις προτάσεις Καρή Μαντελή από τους Πράσινους ως επιτοπλίστων. Στο Συμβούλιο σημειώνουμε ότι θα υπέλθει συμφωνία για το σημείο αυτό εκτός από πλευράς των Γερμανών και των Άγγλων. Ε, με τον ίδιο τρόπο γίνεται μία προστίκη της τροπολογίας 116 που αναφέρει συγκεκριμένα ποια είναι η κατάσταση των εγγύων ε, που ε, αναγκάζονται να εκτεθούν σε αυτό το κίνδυνο. Τέσσερις πολιτικές ομάδες μπορούν να συνυπογράψουν αυτήν την συμβαστική N. περνάμε στην επόμενη O. Ε, επαναλαμβάνουμε τις ε, προτάσεις του σχεδίου γνωμοδότης που είχα προετοιμάσει, δηλαδή ενσωματώνω την νομική υποχρέωση εδώ και τέσσερις πολιτικές ομάδες, ε, έλξοσιαλιστές σοσιαλιστές, και πράσινοι την υποστηρίζουν. Συμβαστική πι εδώ ενσωματώνουμε το θέμα του σεβασμού των πρακτικών ε, και των οικείων πρακτικών και της οικίας νομοθεσίας. Έλξ ε, σοσιαλιστές, φιλελεύθεροι, πράσινοι και συντηρητικοί ικανοποιήθηκαν με αυτή τη συμβαστική. Q. Εδώ επαναλαμβάνουμε τις ε, τροπολογίες 158 και 159 των συναδέλφων Εσάγια και Ντελή και κατά πάσα πιθανότητα σύσσωμες πολιτικές ομάδες την υποστηρίζουν. Για την ε, R, συμβαστική τροπολογία R, μιλάμε για τα κατάλληλα πρότυπα και οι ίδιες πέντε πολιτικές ομάδες δίνουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμβαστική S υπάρχουν ιδέες των σοσιαλιστών σε σχέση με το, τις ε, πρακτικές πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται βάσει της αρχής των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Υπάρχει στήριξη από όλες τις ομάδες. Ταυτόρα, Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγηση αποτελεσματικότητα αυτή τη οδηγία, ε, περιορίζοντα την εφαρμογή στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ε, και ορίζουμε την ε, πενταετία μετά τη θέση εφαρμογή τη οδηγία ω καταληκτική προθεσμία. Επιθυμούμε την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτή τη οδηγία. Τέσσερι πολιτικέ ομάδε ικανοποιήθηκαν με αυτή. ΕΛΚ, Φιλελεύθερη Πράσινη και Συντηρητική. Για τα παραρτήματα, τα αναδιατυπώσαμε, πρόκειται για τι συμβαστικές ε, UW, και X, πρόκειται για τα πρότυπα ICNIRP, της Διεθνούς Επιτροπής δηλαδή για την προστασία από τις σε ακτινοβολίες και μετά τις ε, πληροφορίες του καθηγητή Ζοπελά έχουμε και τη νέα τροπολογία EX, όπου επαναλαμβάνονται οι τροπολογίες 38 και 39 από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και ε, διαγράφοντας επίσης το παράρτημα 4 που είναι άτοπο πλέον διότι έχει ενσωματωθεί ως προς το περιεχόμενό του στα αναδιοτυπωμένα προγενέστερα παραρτήματα. Πέντε πολιτικές ομάδες ε, έχουν δώσει σύμφωνη γνώμη. Θέλω να τονίσω ότι οι εργασίες των πέντε πολιτικών ομάδων με την ενεργό συμμετοχή των σκιωδών ε, εισηγητών οδήγησε σε αυτά τα αποτελέσματα. Είμαι στη διάθεση όλων ε, για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, και με την με κάθε καλή πρόθεση για να, κατα... να υποβάλω και άλλες συμβαστικές τροπολογίες. Κύριε Σιλβάνα Ράπτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, το θέμα αυτό, το εργαζόμαστε πάνω, αυτό, σε αυτό το θέμα πάρα πάρα πολύ καιρό. Ε, θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά την καλή συνάδελφο κυρία Μωρίν Σαρτιέ γιατί ε, κάνει πολύ σκληρή δουλειά και παρά το γεγονός ότι ευχαρίστησε και εκείνη με τη σειρά της του Σκιώδης, η αλήθεια είναι ότι ε, εκείνη χτίζει το σκελετό που είναι το πιο δύσκολο πράγμα Ε, κυρία Πρόεδρε, ξαναρχίζω. Είχα αρχίσει και τα έλεγα πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα τα ξαναπώ από την αρχή. Λοιπόν, ε, ευχαριστώ, λέω, την κυρία Σαρτιέ, γιατί κακά τα ψέματα. Μας ευχαρίστησε όλους τους σκιώδεις συζητητές, αλλά η αλήθεια είναι ότι εκείνη ως εισηγήτρια χτίζει το σκελετό που πρέπει να είναι πάρα πολύ στέρεος και εμείς πάνω σε αυτό βάζουμε πινελιές. Άρα ε, κάνει μια πολύ πολύ δύσκολη ε, δουλειά. Παρακολουθώντας την να αναπτύσσει για μια ακόμη φορά το θέμα των τροπολογιών και των συμβιβαστικών, ε, έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα μελλοντικό γιατρό και αισθάνομαι ασφάλεια πάνω σε αυτό. Λοιπόν, όντως ξεκινήσαμε ε, από άλλες αφετηρίες ενδεχομένως, έχοντας όμως κοινό σκοπό. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι τώρα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε ένα συνενετικό κείμενο. Ε, υπάρχουν ακόμη κάποια ζητήματα. Ε, γι' αυτό και κουβεντιάζουμε βεβαίως ακόμη. Κεφαλαιόδου σημασίας για εμάς, για τους σοσιαλιστές, είναι το ζήτημα των άμεσων και μακροχρόνιων επιπτώσεων στην υγεία των εργαζομένων από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επαρκείς επιστημονικές μελέτες μέχρι τώρα δεν υπάρχουν που να επιβεβαιώνουν τις επιπτώσεις από τη μακροχρόνια έκθεση. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς το ζήτημα. Θεωρούμε επίσης ότι οι έρευνες πρέπει να συνεχιστούν και νομίζουμε ότι κάθε πέντε χρόνια θα πρέπει να εξετάζουμε εάν με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία που καλύπτει τις επιπτώσεις. Προς το παρόν θα πρέπει να έχουμε μία βάση προστασίας που θα παρέχεται από την οδηγία πλαίσιο του 1989. Για τις εξαιρέσεις. Είμαστε σύμφωνοι για τις εξαιρέσεις που υπάρχουν Αξονική τομογράφη και κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις με επιπλέον πρόληψη, με επιπλέον προστασία καθώς και με παροχή σαφών οδηγιών για τον χειρισμό των μηχανημάτων. Ένα άλλο ζήτημα που νομίζω ότι πρέπει ακόμη να εργαστούμε πάνω σε αυτό λιγάκι είναι το ζήτημα ανάμεσα σε οριακές, στις οριακές τιμές έκθεσης, στις ε, exposure limit values και στις τιμές δράσης, action values. Ε, αυτό θα το δούμε λιγάκι ακόμη στην πολιτική μας ομάδα και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι τις επόμενες μέρες να καταλήξουμε. Ε, τελειώνω, δεν θέλω να, να, να μακρηγορήσω. Ε, δηλώνοντας για μια ακόμη φορά την πρόθεσή μας να συνεργαστούμε μέσα στο Κοινοβούλιο ώστε να καταλήξουμε με το Συμβούλιο σε κοινέ θέσεις και σε μια συμφωνία που θα είναι η καλύτερη δυνατή ε, για όλους. Και όταν λέω για όλους εννοώ και για τους ασθενείς που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη το MRI αλλά και για όλους τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά την Μωρίν ε, Σαρτιέ και είμαι εδώ για να εργαστούμε, για να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Alors, euh... Κυρία Μαριάν Άρκιν πρώτα να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την ε, ε, πληρέστη τη γνωμοδότηση και εργασία της και τη διαθέσιμότητά της ε, με πραγματικά εισακούει τις εισηγήσεις των σκιωδών. Ε, για την ε, στις συμβαστικές I and H θα ήθελα να την ευχαριστήσω διότι κάλυψε τις ανησυχίες μας για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Άκουσα μόλις είπε η κυρία Ράπτη ότι έχει κάποια εκκρεμή ζητήματα προς διευκρίνηση για αυτό το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον ε, το ότι συμπεριλάβαμε μέσα συμβαστική τροπολογία το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να επιτείνουν τις προσπάθειές τους για την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων για τις μακροχρόνιες, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ε, ούτως μέχρι ότου να έχουμε διαθέσιμα καταλητικά επιστημονικά στοιχεία και να υπολογίσουμε τις νέες τιμές έκθεση, τότε υποχρεούται, μέχρι τότε μάλλον υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει προετοιμάσει και την αντίστοιχη πρόταση, νέα πρόταση πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Πρέπει να βασιστούμε σε νέα επιστημονικά δεδομένα και η αρχή πρόληψη λαμβάνεται δεόντω υπόψη σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία, κατά τη γνώμη μα. Η συγγήτρια μα μίλησε επίση για το επίθετο biophysical, αν θα συμπεριληφθεί ή όχι. Είχαμε εκφράσει κάποιε ανησυχίε ω προ τη διαγραφή του όρου, αλλά ενδεχομένω να μπορέσουμε τελικά να το δεχτούμε και να αφήσουμε ε, το κείμενο ε, στη μορφή του πιο γενικόλογη, δηλαδή ότι τα τωρινά μέτρα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση όλων των γνωστών ε, επιπτώσεων και να αφήσουμε τον biophysical απ' έξω, αλλά και πάλι ε, ε, ενισχύεται το κείμενο αυτό και ενισχύεται και η προστασία των εργαζομένων. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια διάκριση. Την ίδια την αρχή την ε, επεκτείνουμε και στη συμβαστική Β, όπου μιλάμε για τι ελάχιστε ε, προποθέσει. Ταυτόχρονα λέμε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εναλλακτική λύση να υιοθετήσουν και ευνοικότερε διατάξει εάν το επιθυμούν, στη συμβαστική G ενισχύουμε τις πράξεις εξουσιοδότηση εξασφαλίζοντα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Υγεία και την Ασφάλεια στον χώρο εργασία. Μία ερώτηση ήθελα να απευθύνω για την συμβαστική Q ε, προς την εισηγήτρια. Χαίρομαι που ενσωματώσατε και το νέο κείμενο. Θα ήθελα όμως ε, να σας ε, ζητήσω το εξής. Έχοντας επαναλάβει τώρα το αρχικό κείμενο, ή μάλλον το νέο κείμενο, τι γίνεται με την με τα ε, ε, εντοπιστέντα όρια έκθεσης. Δηλαδή λέμε ότι ο εργοδότης μεριμνά ούτω ώστε η κατάλληλη ιατρική υποστήριξη ε, παρέχεται στους εν λόγω εργαζομένους βάσει του διεθνούς δικαίου και των διεθνών πρακτικών. Αυτό σημαίνει ότι καταπίπτει το υπόλοιπο κείμενο κατά τη γνώμη μας διότι λέει στη συνέχεια ότι το κόστος θα πρέπει να το φέρει ο εργοδότης αλλά είναι προφανές ότι αν ο εργοδότης πρέπει να μεριμνά ούτως ώστε να παράσχει το κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό νομίζω ότι πρόκειται για επανάληψη και είναι περίτω. Στη συνέχεια λέμε shall be performed, θα γίνεται σε ώρα, εν ώρα εργασίας. Ε, ενδεχομένως αυτό να μην ε, ικανοποιεί τον εργαζόμενο. Οπότε να το συζητήσουμε σύντομα δεν είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα να καταλήξουμε σε συμφωνία και με πολύ λίγη συζήτηση. Επίσης, ε, για όλους όσους ανησυχούν ακόμη για την υγεία των εργαζομένων, ενισχύσαμε και τη συμβαστική ΕΜΕ, εισαγάγοντας το, την εξή αράδο εργοδότης, έχει την υποχρέωση και θα αναλάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ότι ο κίνδυνος προέρχεται από την έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στο χώρο εργασίας, ε, απαλήφεται ή περιορίζεται στο ελάχιστο. Ε, θα έχουμε εργαστεί πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ σημαντική η γνωμοδότηση και είναι και και σημασία να συνεχίσουμε τα περί μαγνητικής τομογραφίας, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν εκεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε πάρα πολλά άλλα ζητήματα, εξαιρετικά τεχνικά, κυρίως μέσα στα παραρτήματα. Ε, πάντως χρησιμοποιούμε τις ε, πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες και θα βασιστούμε στα, στις πληροφορίες που μας δίνει η ΙΚΝΕΡΠ. Πιστεύω ότι στο Συμβούλιο θα καταστεί δυνατόν να ε, κλείσουμε μία συμφωνία. Ήταν επικοδομητική και ε, πληρέστατη η εργασία μας και η συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Μακιντάι. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Ελίζα για την πολύ σκληρή δουλειά που κατέβαλε. Πιστεύω ότι σταδιακά έχουμε καταφέρει να συμφωνήσουμε με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Την ευχαριστώ λοιπόν για αυτό. Υποστηρίζω πολύ, ουσιαστικά οτιδήποτε κάνει. Ο τομέας που μας απασχολούσε περισσότερο, όπως και κάποιους άλλους, είναι τα μακροπροθέσμα αποτελέσματα για την υγεία και πιστεύω ότι δεν πρέπει να προσπαθούμε να προδικάσουμε τα αποτελέσματα μελλοντικών ερευνών. Υποστηρίζουμε δηλαδή τη συνέχιση των ερευνών περαιτέρω επιστημονικών ερευνών για τις ε, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να υπερασπίσουμε τροπολογίες που προδικάζουν τα αποτελέσματα πριν μάθουμε τα αποτελέσματα των ερευνών αυτά. Αλλά πιστεύω ότι όλες αυτές οι τροπολογίες και οι συμβιβασμοί ε, συντείνουν σιγά σιγά και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την κυρία Μορασάρτια για το έργο της ε, Πρόεδρος Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω δει καθόλου αυτό το φάκελο. Σας εμπιστεύουμε όλου, αλλά καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, με απασχολεί η δυναμική την οποία θετούμε Το ερώτημα εν τέλει είναι να δούμε πώς λαμβάνουμε υπόψη ε, την εξέλιξη της γνώσης των επιστημών και το πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τους ασθενείς, τους εργαζόμενους και τον εξοπλισμό. Εγώ καταλαβαίνω ότι τα όσα έχουν υλοποιηθεί από την ομάδα ε, επιτρέπουν ουσιαστικά να υπάρχουν κατεξούδα της πράξης. Μια επισκόπηση του τι μπορεί να τροποποιήσουν ή να συμπεριλάβουν οι κατεξούδα της ε, στην ίδια την οδηγία και ένα αίτημα για μια οδηγία για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Εγώ απλά θέλω να είμαι βέβαιη ότι με αυτό το μέσο θα καταλήξουμε σε μια οδηγία στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι προόδοι της έρευνας και της ανάπτυξης τόσο όσον αφορά τον νέο εξοπλισμό διότι διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος κάποιοι υπεύθυνοι για μηχανική τομογραφία να μου πούν δεν μπορώ να εφαρμόσω τα δικά σας πρότυπα διότι τα δικά μηχανήματα είναι πιο ασφαλή Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιπτώσεις της μαγνητικής τομογραφίας για τους εργαζομένους ε, και δεν θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις λόγω των δικών μας νομοθετημάτων. Θέλω λοιπόν να ξέρω το πεδίο που καλύπτουμε με τις κατεξουδότησης πράξεις και την επισκόπηση των κατεξουδότησης πράξεων να μπορούμε να καλύψουμε όλο αυτό το πεδίο εφαρμογής διότι όπως γνωρίζετε ήταν δύσκολο να καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν θα παγώσουν όλα ε, ή θα απομονωθούν ουσιαστικά διότι δεν είναι πλέον εφαρμόσιμα λόγω εθνικής νομοθεσίας. Ο κύριε Σίλβα το πρωί σήμερα είναι δικό σας και μετά η κυρία Συγγήτρια. Κύριε Σίλβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην παρουσιαφάση δεδομένου ότι τα τελευταία κείμενα των τροπολογιών ε, μας είναι πλέον γνωστά Δεν θα κάνω σχόλια. Χρειάζεται πρώτα κάποια μελέτη. Σίγουρα θέλω και εγώ να συγχαρώ όπως και οι υπόλοιποι την κυρία Συγήτρια για την δουλειά της η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και ελπίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να καταλήξουν σε ε, συμβιβασμού τηρώντα τις πολύ μας προθεσμίες. Θα ήθελα απλά να πω δύο λόγια για να εκφράσω μια επιφύλαξη όσον αφορά μία από τις τροπολογίες που προβλέπονται σε αυτό το κείμενο. Αφορά την υποχρέωση προς την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση ε, οδηγίας σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των ερευνών. Σας υπενθυμίζω ότι η οδηγία, η εν λόγω οδηγία, θα εγκριθεί βάσει του άρθρου 153, το οποίο έχει σκοπό τον ορισμό υποχρεώσεων για τα κράτη-μέλη. Η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να μεταφερθεί στην Εθνική Νομοθεσία από τα κράτη-μέλη. Μια οδηγία βάσει του άρθρου 153 δεν έχει σκοπό να επιβάλλει υποχρεώσει στην Κομισιόν. Η Κομισιόν πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα πρωτοβουλία τη και μάλιστα αν μιλάμε για ερευνητικά προγράμματα πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι αυτή η διάταξη θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό την οδηγία. Αλλά για έρευνα της Κομισιόν υπάρχουν άλλα μέσα. Δηλαδή οι γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου είναι πιο κατάλληλες για αυτό το σκοπό. Σας ε, δηλώνω λοιπόν μια επιφύλαξη εκ μέρους της Κομισιόν για αυτό το σημείο, αλλά σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε πιο λεπτομερώς στο μέλλον. Ευχαριστώ. Δεν ε, μπορώ να αντισταθώ να... στον αντιδράσω σε αυτό που λέτε με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής. Είμαστε οι πρώτοι που θα πούμε ότι η Επιτροπή καταχράται τις δυνατότητες που έχει να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς σίγουρα θα υπάρχουν κάποιες ε, διευθετήσεις. Φυσικά θα το κοιτάξουμε με το όλη τη ε, με το δέον ζήλο. Έχουμε το άρθρο 153 της συνθήκης και δεν είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα σας επιβάλλω την ανάγνωση όλου του κειμένου που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας. Νομίζω όμως ότι μπορούμε, ε, θα μπορέσουμε στα πλαίσια τα σημερινά να έχουμε μια σωστή σύνταξη κειμένου και να σεβαστούμε την, ε, την νομική βάση. Θα δώσω όμως το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Σαρτιέ τώρα. Έλαβα υπόψη τις παρατηρήσεις που γίνανε από όλου τους συναδέλφους και σιωδησίτες. Θα ήθελα να πω ότι παρόλο που έλειπε η Καρυμαντελή σήμερα το πρωί, δεν μπορούσα να είναι παρούσα, μετά από μεγάλη συζήτηση με το σκιώδη κυρίως για το θέμα του όρου biophysics, φαίνεται ότι η Κάρη Μαντελή, εκ ονόματος των Πρασίνων, θα συμφωνούσε να διατηρήσουμε την διευκρίνηση, την ακρίβεια αυτού του όρου στον ορισμό που δίνουμε, σε αντίθεση με την ε, τελευταία συζήτηση που είχαμε κάνει. Θα πρέπει να το, ε, επανα, να το ξαναπούμε στους συναδέλφους από από τους φιλελεύθερου, γιατί συζητήθηκε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσω απλώς. Συγκυρία Ράπτη τώρα, για την αναθεώρηση, για την ε, επανεξέταση κάθε πέντε χρόνια αυτή εδώ τη οδηγία. Είχαμε συζητήσει, αγαπητή Σιλβάνα, πάρα πολύ, κυρίως στην τελευταία συνεδρίαση με τη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών και είχαμε πει ότι αυτό, αν είχαμε αυτό το θέμα έτσι, αυτό θα απέβαινε εις βάρος του συμφερόντων των εργαζομένων, διότι ότι από τη στιγμή που υπάρχει, υπάρχει πληροφόρηση για, τα ενδεχόμενα, για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, θα πρέπει τότε να δούμε να αναθεωρήσουμε την οδηγία. Αν περιμένουμε πέντε χρόνια, ξέροντας φέρει πίνο ότι για τέσσερα χρόνια υπάρχουν ε, ενδυνάμει αρνητικές επιπτώσεις, τι κάνουμε. Κανένας δεν θα είχε ήσυχη τη συνείδησή του. Γι' αυτό λοιπόν προτιμήσαμε αυτή την απανδραστηριοποίηση, διότι δε μη θα είχαμε μεγάλα κενά σε σχέση με το θέμα της υγείας των εργαζομένων σε επιπτώσεις μπορούν να έχουν από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσω διότι έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και έχουμε προβληματιστεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα με τους εμπειρογνώμενες, με τους χρήστες, με τους ε, ασθενείς, με τις διάφορες πολιτικές ομάδες και καταλήξαμε ότι αυτή είναι η θέση η σωστή και την οποία ειλικρινά θα θεωρώ ότι έπρεπε να τη διευκρινίσω για τον όρο Biophysics. Ε, μίλησα ειδικά με τη Μαριάν Αρκίν σε σχέση με την ε, θέση των Πρασίνων. σας ευχαριστώ την κυρία Μακεντάιρ που μου δείχνει εμπιστοσύνη και σε εσά τώρα κυρία Πρόεδρε. Άκουσα τις παρατηρήσεις, την παρατήρησή σας Έκαναμε μια συνάντηση σημαντική που μας πρόσφερε πάρα, πολύ, πάρα πολλές διευκρινήσεις ΠΑΚ. Με την ενότητα, στη, με υπερογνώμονες ειδικού στο Στρασβούρ έγινε αυτό. Έχουμε την συνάδελφο Ανταλής Γκρισμπεργκ που ήταν μαζί μας και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Είχαν έρθει αυτοί όμως. Πιστεύω ε, πραγματικά ήταν πραγματικά το νόημα της εργασίας μας να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των της ε, μαγνητικής ομογραφίας και απ' την άλλη να έχουμε την προστασία των εργαζομένων. Εμείς πραγματικά μπήκαμε στη θέση ε, αυτών για να δούμε το θέμα της προστασίας των εργαζομένων. Σήμερα το κείμενο που σας προτείνεται και οι συμβαστικές προτάσεις λαμβάνουν υπόψη αυτή τη διπλή ισορροπία. Δεν είναι... Δεν ε, έχουν να κάνουν με τις μελλοντικές, μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά τον εξοπλισμό. Σήμερα αυτό που βλέπουμε ότι προσπαθεί κανείς όσο δυνατόν να μειώσει το, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και προσπαθεί να εξασφαλίσει τις καλύτερες και πιο ασφαλείς συνθήκες. Το κείμενο λοιπόν όπως σας, προτείνετε σας το προτείνουμε σήμερα λαμβάνει υπόψη στο σύνολο αυτές τις πτυχές. Και με αυτόν τον τρόπο απαντάω στην παρατήρηση τη Επιτροπής. Όντως η Επιτροπή ε, θα πρέπει να βάλει τα δυνατά της και να μας ε, βοηθήσει να δουλέψει ούτω ώστε να μπορούμε να έχουμε εφαρμογή αυτής, μέσα σε πλαίσιο 5 ετών αυτής της οδηγίας στις χώρες μέλη. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει αποδεκτό να μην πρέπει να έχουμε την εφαρμογή ταυτόχρονα με την παρακολούθηση της επιστημονικής εξέλιξης. Δηλαδή μια διτή δέσμευση. Είναι πολύ σημαντικό κατά με να επιμείνουμε σε αυτό. Ξέρουμε ότι και εδώ θα πρέπει στη συνεργασία με το Συμβούλιο να έχουμε σημαντικές και αυστηρές ε, συζητήσεις. Είμαστε έτοιμοι. η σύγκληση τώρα ε, απόψεων διαφόρων πολιτικών ομάδων που ήταν διαφορετικές αλλά σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνένεση δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο. Όλες οι πολιτικές ομάδες ε, εντάσσονται σε αυτές τις βασικές προτάσεις. Βλέπουμε δηλαδή τη θέληση που υπάρχει να δούμε τα, το ρίσκο μακροπρόθεσμα από τη μια και από την άλλη η, τη δέσμευση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας κάθε πέντε χρόνια για την εφαρμογή της. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα καταχραστώ τις θέσεις μου ως πρόεδρος για να σας κάνω μια μικρή ερώτηση. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι, εντάξει, για τους εργαζόμενους κατάλαβα ότι καλύπτονται, ότι αν ξαφνικά ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν παρενέργειες, ε, έχει προβλεφθεί αυτό. Ο άλλο κίνδυνος όμως στην αντίθετη κατεύθυνση είναι ότι η βιομηχανία ξαφνικά μπορεί να ανακαλύψει ένα εξαιρετικά αποδοτικό μηχάνημα το οποίο επιτρέπει ε, μαγνητική τομογραφία με χαμηλότερες, ε, χαμηλότερη ακτινοβολία και ξαφνικά λένε α, τη σκίζουμε αυτή την οδηγία γιατί δεν έχει πλέον εφαρμογή. Αυτό με ενδιαφέρει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν μιλάμε για ακτινοβολία φυσικά, διότι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επιτρέπουν να μην χρησιμοποιούνται ακτινοβολίες οι, οποίες αυτές είναι επιβλαβείς, ενώ σήμερα τα μαγνητικά πεδία δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι είναι επιβλαβή. Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια εφαρμογής αυτής της, ε, την εφαρμοσιμότητα θα έλεγα αυτής της οδηγίας ε, σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις προόδους ε. καμία επίπτωση σήμερα δεν θα επέτρεπε να καταστεί άκυρη αυτή η οδηγία διότι πρόκειται για διεθνή πρότυπα. Όλα τα μηχανήματα ούτως ή άλλως πρέπει να τηρούν αυτά τα διεθνή πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα και στα παραρτήματα. Πρέπει να σας πω κυρία Πρόεδρε ότι παρότι η δυσκολία του έργου μας ε, μεταξύ των πολιτικών ομάδων, επειδή υπήρχε καλή θέληση από όλα τα μέρη, τα πράγματα δεν ήταν τόσο δύσκολα. Οι δυσκολίες ήταν η συνεργασία με το Συμβούλιο, διότι ακριβώς τα παραρτήματα για το εν λόγω πρόβλημα ε, άρχισαν να γίνονται τεράστια και η Προεδρία του Συμβουλίου ξεκινούσε να συζητά πάντα ορισμένες φορές από τα παραρτήματα, άλλες φορές από το κείμενο, τα εξετάσαμε, τα επανεξετάσαμε, προσπαθήσαμε να τα ε, δουλέψουμε κάπως. Ε, πιστεύουμε ότι καταλήξαμε σε κάτι εποφελές για τους εργαζόμενους, για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, για την υγεία των εργαζομένων ενώ και για τους ασθενείς. Πραγματικά θα ήθελα πολύ ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές από τις διάφορες πολιτικές ομάδες καθώς και τη γραμματεία της Επιτροπής μας που ήταν πάντα στη διάθεσή μου και βοήθησε εξαιρετικά και θα ήθελα ειδικότερα να ευχαριστήσω τον κύριο Ερμπίγιου από την Επιτροπή που για πολύ καιρό ήταν μαζί μας και συνεργάστηκε μαζί μας επί του θέματος. Ευχαριστώ. Πολύ καλά λοιπόν βάσει αυτής της συζήτησης με τις τόσες πληροφορίες που ακούσαμε θα ψηφίσουμε στις 6 Δεκεμβρίου και μετά θα περάσουμε στη μεγάλη διαπραγμάτευση που από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι λιγότερο περίπλοκη. Μας απομένει ένα θέμα. Προχωράμε σιγά σιγά τα πράγματα. Έχουμε το σημείο 16. Κυρία Μωρανσαρτία, σας ξαναδίνω το λόγο για να μας παρουσιάσετε την τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο στο πλαίσιο του τριμερούς διάλογου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κυρία Ισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να πρωτοπώ από αυτές τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Το είπατε κι εσείς, ήταν πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του τριμερούς αυτού διαλόγου. Ε, οφείλω να πω ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει ένα ρόλο ε, εξισορροπητικό και ευεργετικό θα έλεγα, διότι το Συμβούλιο ακόμη δεν έχει διαπραγματευτική εντολή ξεκάθαρη. Καθυστερεί για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα χρειάστηκε να συμφωνήσουμε ε, για τη μεθοδολογία εργασίας. Δόξα το Θεό είναι και το ατού μας αυτό, διότι στα πλαίσια του διαλόγου αυτό ατού είναι η έκβαση της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Απασχόλησης, χάρη στην οποία από πλευράς Κοινοβουλίου έχουμε ε, μια ισχυρότατη διαπραγματευτική εντολή. Δεύτερον, η προσήλωση των ε, σκιωδών από πλευράς των διαφορών πολιτικών ομάδων, διότι είναι εξαιρετικά αφοσιωμένοι και προσιλωμένοι όλοι οι σκιώδες επαρκείς, κατέχουν το ζήτημα και θα ε, με ακολουθήσουν όπως και εσείς στις διαπραγματεύσεις ιδιαίτερα αποφασισμένοι να επιτύχουν τους στόχους τους. Επίσης ε, έχουμε ένα άλλο ατού τη γραμματεία μας ε, και ευχαριστώ την κυρία Νιελή και την κυρία Σοντέ γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ από πλευράς της γραμματείας για την για να τα καταφέρουμε. Έχουμε φτάσει στο πέμπτο στάδιο του τριμερούς και δεν έχουμε μόνο την ενεργεία προεδρία ε, που εκπροσωπείται σε αυτές τις ε, συσκέψεις, ε, αλλά εκπροσωπείται και η επερχόμενη Ιρλανδική προεδρία. Και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κυρία Μανουέλα Γκελέγκ από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση προχωρούμε βάσει θεματικών ενωτήτων. Ε, επεξεργαστήκαμε τα άρθρα, ε, υιοθετώντα αυτή την θεματική προσέγγιση και είδαμε κάθε άρθρο ξεχωριστά. Υπάρχουν σοβαρά προσκόμματα ε, και κάθε φορά πρέπει να επιχειρηματολογούμε ε, ακόμη και για προφανή, για προφανέστατα σημεία. Παραδείγματο χάρη για τη δημοσίευση των ε, στοιχείων Bixible, ε, καταφέραμε να βρούμε μία κοινή προσέγγιση για τους ε, νέους για τις ε, επαγγελματικές ε, δεξιότητες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα και καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τριμερή διάλογο έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες και πρέπει να εξετάσουμε μια νέα πρόταση διατύπωσης που ενδεχομένως να τύχει της αποδοχής των ομάδων, αλλά ταυτόχρονα ε, επιχειρηματολογούμε ε, με επιχειρήματα που κανονικά θα έπρεπε να εξεταστούν στο Συμβούλιο Στο μέτρο που δεν υπάρχει διαπραγματευτική εντολή, καθυστερούμε. Καθυστερούμε υπερβολικά διότι δεν έχουμε τη διεπαφή της ε, συζήτησης ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα που θα εξασφάλιζε και την αίσια πορεία των διαπραγματεύσεων και εγώ πραγματικά έχω αμφιβόλειες να επαναλαμβάνονται δηλαδή ε, αδιάκοπα οι τριμερείς αυτοί διάλογοι. Πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα προγραμματισμού που θα πρέπει να εξαγάγουμε στην Επιτροπή. Είναι γεγονός ότι μας περιγράφεται μια κατάσταση που βρίσκουμε, αντιμετωπίζουμε σε πολλοί στριμερείς διαλόγους. Καταλαβαίνει κανείς ότι το ότι δεν έχουμε επιστροφή του έργου μας από την Συμβουλίου έχει να κάνει ότι δεν ε, δεν υπάρχει θέληση βασικά να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα σε νομοθετικό επίπεδο όσο θέλαμε. Σας ευχαριστώ που μας παρουσιάσατε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν κάποιος συνάδελφο θέλει να πει κάτι. Ο συνάδελφος Γκέρο Ροσαλόμ δεν επιθυμεί να πάρει το λόγο και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε για σήμερα και μάλιστα πιο νωρίς. 6 Δεκεμβρίου στην επόμενη συνεδρίαση που θα είναι και πολύ δυναμική.